El señor Επαναλαμβάνονται οι εργασία τη Συνόδου. Τα πρακτικά της προηγούμενης Συνόδου είναι διαθέσιμα και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θεωρούμε ότι εγκρίνονται. Και περνούμε στο σημείο το ακόλουθο της διάταξης που είναι η κοινή συζήτηση για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, χρηματοπιστωτική κρίση και αμυντικός τομέας. Έχουμε την δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και υπάτης εκπροσώπου της Ένωσης, της κυρίας Άστον, και έχουμε και την έκθεση ΛΙΣΕΚ για τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον αμυντικό τομέα. Όπως είπα, πρόκειται για κοινή συζήτηση. Η κυρία Άστον έχει το λόγο. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Λίσεκ για την έκθεσή του. Όπως είπα χθε το βράδυ που τον συνάντησα, Ήμουν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας ε, και μου είπαν ότι ε, θέλουν να διαβιβάσω στον εισηγητή τι ευχαριστίες τους για το έργο του. Φυσικά σε ό,τι αφορά ε, την ε, συζήτηση για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ε, της οικονομικής κρίσης που οδήγησε σε μεγαλύτερη εστίαση στην συγκέντρωση και κοινή χρήση των αμυντικών δυνατοτήτων και στις ελλείψεις προσωπικού, κάτι το οποίο βλέπουμε σε διάφορες σημαντικές επιχειρήσεις και αποστολές της ΕΠΑ. Πρέπει λοιπόν να τα κάνουμε καλύτερα τα πράγματα και έστω και με τους λιγότερους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι πολύπλοκη κατάσταση, έχουμε την κρίση, έχουμε τις κυβερνοεπιθέσεις, την ενεργειακή ε, κρίση και πολλά άλλα. Πολλές άλλες προκλήσεις. Πρέπει επίσης ε, να είμαστε αποδοτικοί ε, μέσα στο οικονομικό πλαίσιο που έχουμε και θα πρέπει οι δράσεις της ΕΠΑ να βασίζονται σε Συνεκτικέ δράσει σε μια παγκόσμια συνολική προσέγγιση και βέβαια θα πρέπει να είμαστε εξοπλισμένοι με τι ε, απαραίτητε δυνατότητε, όπω υπόθηκε και την 1η Δεκεμβρίου στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Έχουμε δημοσιονομικού περιορισμού, άρα πρέπει να εξοικονομήσουμε πόρου, αλλά συγχρόνω να έχουμε στενότερη συνεργασία. Είτε με τη συγκέντρωση και κοινή χρήση των πόρων, το κοινό πρόγραμμα τη αναπτυξιακή βοήθεια, αλληλεγγύη σε ό,τι αφορά την ε, κένωση, την απομάκρυνση Ευρωπαίων πολιτών από περιοχέ που βρίσκονται σε πόλεμη κατάσταση κατάσταση ή ε, υπάρχει κάποια έκτακτη ανάγκη. Επίση, ε, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων εγκρίθηκε η δική μου έκκληση να έχουμε μεγαλύτερε συνέργειε και ε, να μην αλληλοκαλυπτόμαστε αλλά να αλληλοσυμπληρωνόμαστε η δράση επίσης που θα αναλάβει η εξωτερική, υπηρεσία εξωτερικής δράσης και η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, αλληλοενισχύονται. Στη συνεδρίαση της 1 η Δεκεμβρίου επίσης συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να βελτιώσει τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκή Ένωση προσδιορίζοντας με σαφήνεια τις ανάγκες και ε, βρώντας με σαφή στόχους ε, και στρατηγικές εξόδου μαζί με τα Εθνικά Κοινοβούλια και τι κυβερνήσει, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο για να υπάρχει δημοκρατική εποπτεία και έλεγχος ε, τη εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνα και ασφάλεια. Το έχω πει και στη δήλωσή μου για την πολιτική ευθύνη. Θα ήθελα τώρα να επικεντρωθώ σε κάποιες από, ε, από τα σημαντικά επιτεύγματα τη τελευταία χρονιά στο τομέα των δομών. Έχουμε την ΕΙΕΔ πλέον, η οποία πλέον είναι εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει καλύτερα, ταχύτερα και ευφιέστερα τις κρίσεις. Όταν Λοιπόν, δρομολογήθηκε η υπηρεσία αυτή τον Ιανουάριο 2011, απαιτούσε την άμεση αντίδρασή μα η Αραβική Άνοιξη. Και με βάση τι εμπειρίε μα, συγκροτήσαμε το Συμβούλιο Διαχείριση Κρίσεων και την πλατφόρμα τη ε, κρίση, που επίση ε, αντιμετώπισε πολύ επιτυχημένα καταστάσει κρίση ε, στην ακτή Ελεφαντοστού, τη Λιβύη και το κέρα Αφρική. Και είναι σημαντικέ αυτέ οι δομέ για τη δυνατότητα που έχουμε να αντιδράσουμε, αλλά και να συνεργαστούμε ε, ε, βέβαια με την υπόλοιπη υπηρεσία, αλλά εγώ πρέπει να διατηρώ τη βασική ευθύνη. Επίσης βελτιώσαμε και την, ε, το μέσο έγκαιρης προειδοποίησης ε, με την ομάδα για την πρόληψη των συγκρούσεων και το λεγόμενο Situation Room και θα δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις, την εμπειρογνωμοσύνη μας στις αντιπροσωπείες και ε, όλα αυτά τα κάναμε με την αναδιάρθρωση των υφιστάμενων ε, πόρων ε, και βελτιώντα την ευελιξία, την αποτελεσματικότητα αυτών, χωρί να αναζητήσουμε δαπανηρέ πολύπλοκε λύσει. Αυτό το οποίο πλέον πρέπει να κάνουμε είναι μια συλλογική συνεκτική προσέγγιση και να την μετατρέψουμε σε δράση. Και είμαστε με την ΕΙΕΔ, νομίζω έχουμε τα κατάλληλα μέσα στη διάθεσή μας, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, να προλάβουμε κρίσεις και αυτή την ε, υπηρεσία θα τη θέσουμε ε, στην υπηρεσία ε, της Ένωσης για την αντιμετώπιση κατάστασης στο τη Αφρικής και στην Νότια Γειτονία. Κάποιοι λένε ότι υπάρχει ένα είδος κόπωσης με την ΚΕΠΑ, αλλά θα έλεγα αντίθετο το 2011 ήταν ένα έργο εντατικής δουλειάς με πολύ απτά αποτελέσματα και η κατάληξη ήταν κάποια συμπεράσματα του Συμβουλίου τα οποία θα τα χαρακτήριζα πλήρη ε, και κοιτώντα προ το μέλλον. Τότε θα στρατιωτικέ δυνατότητε. Έχουμε την Συντονιστική Επιτροπή του Οργανισμού Άμυνα που έδωσε συγκεκριμένε δεσμεύσει σε συγκεκριμένα σχέδια όπω σε τομεί που είδαμε ότι υπάρχουν ελλείψει, όπω με την κρίση τη ε, Λιβύη και θα παραστώ επίση ε, και την άνοιξη την επόμενη στο σε διάσκεψη κορυφή του ΝΑΤΟ στο Σικάγο. Και στην έκθεση λύση εκλέγεται ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία. Η πολυεθνική συνεργασία πρέπει να γίνει κανόνα και όχι να είναι η εξαίρεση, αν θέλουμε να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε τι αμυντικέ δυνατότητε τη Ευρώπη. Συμφωνώ με αυτό το οποίο λέει ο κύριο Λίσικ, δηλαδή ότι η συγκέντρωση και κοινή χρήση πόρων, το pooling and sharing, είναι ένα τρόπο να έχουμε και βελτιωμένε δυνατότητε και να αντιμετωπίζουμε επαρκώ. Ε, τι περικοπές στου αμυντικού προπολογισμού. Ως επικεφαλής ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνα, θα συνεχίσω να καταβάλω κάθε προσπάθεια για να υπάρχει εύκολη, καλή συνεργασία μεταξύ, και, ε, μεταξύ των κρατών μελών και για να υπάρξει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα στην αμυντική βιομηχανία. Τον Ιούλιο παρουσίασα μία έκθεση για την ΚΕΠΑ και εκεί ανέφερα τι παραμέτρου και για την περαιτέρω εργασία και σε ό,τι αφορά το hardware και το software, αφενό δηλαδή στρατιωτικέ και μη στρατιωτικέ δυνατότητε και αφετέρου πώ θα σχεδιάσουμε και πώ θα συνεργαστούμε με του εταίρου μα. Και ε, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων τη 1η Δεκεμβρίου χαιρέτησε το σχετικό μου έργο. Οι πρωτοβουλίε των κρατών μελών, όπω είναι η πρωτοβουλία τη Βαϊμάρη ε, και άλλε συμβολέ, νομίζω ότι έχουν δώσει περαιτέρω όθηση στι εργασίε μα. Επίση, χαίρομαι γιατί βρήκαμε έναν αρελιστικό τρόπο να προχωρήσουμε ε, σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων ΚΕΠΑ και θα έχουμε τώρα και το κέντρο ε, επιχειρήσεων για όλες τις επιχειρήσεις στην Αφρική που θα το εγκρίνουμε τον Ιανουάριο στο επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και έτσι θα μπορέσουμε να δούμε αν λειτουργεί καλά ε, αυτό το εργαλείο γιατί θέλουμε να ενθαρρύνουμε την ενδυνάμωση των ε, συνεργειών στρατιωτικών και μη στρατιωτικών μέσων και να κλείσουμε διδάγματα για το μέλλον. Νομίζω ότι με τη συνεργασία μα με του εταίρου έχουμε καταφέρει σημαντική πρόοδο. Στον τομέα τώρα τη ασφάλεια και τη άμυνα, η σχέση με τον ΝΑΤΟ είναι σημαντική και αναγνωρίζεται και στη συνθήκη τη Λισαβόνα. Την πρώτη από τι ε, συνθήκε τη Ένωση που αναφέρεται ρητά ε, στο ΝΑΤΟ. Θα μπορούσαν λοιπόν όλο το φάσμα από των εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνδυαστούν με τον πολύ σημαντικό ρόλο που έχει το ΝΑΤΟ για τα αμυντικά θέματα και οι δύο οργανισμοί νομίζω ότι μπορούν από κοινού να αλληλοενισχύσουν τις εργασίες τους. Με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, κύριο Ράσμουσεν, έχουμε συνεργαστεί στενά για να έχουμε μια προσέγγιση βαθμιαία αλλά ρεαλιστική για τη συνεργασία των δύο οργανισμών η κρίση της Λιβύης έδειξε για μια ακόμη φορά ότι αυτό είναι αναγκαίο και πραγματικά σε πολλά θέατρα επιχειρήσεων συνεργαζόμαστε. Αυτό το οφείλουμε ε, στους ανθρώπους μας, ε, στους αριθμούς μας που είναι επιτόπου. Και χαίρομαι που επιβεβαιώνω ότι σε ό,τι αφορά ιδίως τις δυνατότητες ε, Ήδη έχουμε πετύχει έναν ευπροηγουμένο επίπεδο συνεργασία. Είτε το ονομάζει κανεί αυτό εφιάμινα, είτε pooling και sharing. Και τα Ηνωμένα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σταθερό εταίρο. Αυτή την εταιρική σχέση την κάνουμε πλέον την ε, κάνουμε πράξη. Ε, στο Αφγανιστάν, στη Σομαλία, στο Κοσφοπέδιο, στην Λιβύη, εκεί δηλαδή που είμαστε ε, ή θα μπορούσαμε να είμαστε παρόντε ε, στα θέατρα αυτά των επιχειρήσεων ή και μέσω του στρατηγικού διαλόγου. Έχω επίση τονίσει πόσο σημαντική συνεργασία με στρατηγικούς εταίρους και φυσικά βλέπουμε στρατηγικά θέατρα επιχειρήσεων το κέρας Αφρική και τη Λιβύη. Έχω υπογράψει επίσης σύμβαση πλαίσιο με τις ΗΠΑ τον Ιούνιο για τη συμμετοχή τους σε πολιτικές αποστολές και ΕΠΑ. 60 Αμερικανοί ήδη ε, είναι κάτω από τη διοίκηση, την αλυσίδα διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κοσμοπέδιο και το Αφγανιστάν, αλλά θέλω να ενισχύσω τη συνεργασία και με άλλες ε, γειτονικέ χώρες και τις, ε, τους γείτονες προς ε, Ανατολάς και προς Νότον. Ολοκληρώνοντα παρατήρησουμε παρατηρήσει μου, θα να σα μιλήσω για το μέλλον. Πρέπει ε, να είναι πιο επιχειρησιακή αυτή η συνολική προσέγγιση, το comprehensive approach. Θα πρέπει καλύτερα να συσχετίσουμε τι δραστηριότητέ μα στον τομέα τη πρόληψη, τη διαμεσολάβηση, τη ανάπτυξη, τη επίλυση συγκρούσεων. Και βέβαια έχει και, και πολύ σημαντικό ρόλο να ε, διαδραματίσει για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματο, ε, το λαθρεμπόριο όπλων, τα ναρκωτικά και την εμπορία ανθρώπων. Όλα αυτά σχετίζονται με συγκρούσεις, όπως είδαμε και τις ε, απειλές ε, στο Σαχέλ, σε ό,τι αφορά το της ασφάλειας, που έχουν να κάνουν και με τη ροή όπλων και ε, ανταρτών. Πάρα πολύ σημαντική λοιπόν εδώ είναι η δυνατότητα που θα έχουμε να συνδυάσουμε όλα τα εργαλεία της Ένωσης. Επίσης σημαντική και σταθερή πρέπει να είναι η προσοχή μας για την αύξηση των δυνατοτήτων μας ε, και της, ε, την παραγωγή δυνατοφόρτς generation που θα πει οι σωστοί άνθρωποι στο σωστό μέρος. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, στρατιωτικές δυνατότητες θα πρέπει να έχουμε συστηματική συγκέντρωση και κοινή χρήση των πόρων όχι μόνο για να αντιμετωπίσουμε τους οικονομικούς περιορισμούς αλλά για να βελτιώσουμε ε, την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα μακροπρόθεσμα και θα πρέπει και την αποτελεσματικότητα των αποστολών και των επιχειρήσεων να τη βελτιώσουμε. Θα πρέπει μέσω των αποστολών ε, και επιχειρήσεων και ΠΑ να προσπαθεί να δημιουργεί προστιθέμενη αξία βάσει των αναγκών που θα έχουν ε, εντοπιστεί με σαφείς στόχου και στατικές εξόδους. Ό,τι αφορά τώρα τα παραδοτέα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τις εφιστάμενες αποστολές, ιδίως σε πολύ σημαντικές στρατηγικά περιοχές όπως το Σαχέλ και η Λιβύη, θα πρέπει ε, να εργαστούμε και ε, για νέες αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αποτελεσματικοί και φιλόδοξοι στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ, αλλά αυτό βασίζεται σε μια συλλογική πολιτική βούληση και φιλοδοξία. Και σε ό,τι αφορά το προπολογισμό θα πρέπει να είναι κατάλληλο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Και θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξή του σε αυτού του μήνε. Ολοκληρώνοντα, σα ευχαριστώ για την υποστήριξή σα, ό,τι αφορά τι δικέ μου εργασίε για την ΚΕΠΑ. Και θέλω να επανεπιβεβαιώσω, θα συνεχίσω να είμαι δεσμευμένη ε, στην ε, πολιτική αυτή που αποτελεί ένα αναπόσπαστο και πάρα πολύ απαραίτητο τμήμα τη εξωτερική δράση Ευρωπαϊκή Ένωση και ευχαριστώ εκ νέου τον κύριο Λίση για την έκθεσή του. Σα ευχαριστούμε κύριε Άστον. Τώρα για τέσσερα λεπτά θα λάβει τον λόγο ο κύριο Λίσεκ. παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ πρόεδρε είπατε εκπρόσωπε κυρίες και κύριοι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα θερμά λόγια που στόχευαν στην έκθεσή μου. Ήθελα να τονίσω ότι είναι η έκβαση της κοινής, του κοινού μας έργου, όχι μόνο της δικής μου εργασίας, αλλά και πάρα πολλών μελών από διαφορετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές ε, όσον αφορά θέματα άμυνας και ασφάλειας και, θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους σκιώδεις εισηγητές με τους οποίους η συνεργασία ήταν πραγματικά χαρά για μένα. Τους ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία τους. Με μεγάλη ικανοποίηση άκουσα, πρέπει να πω ότι εσείς ε, κυρία είπατε εκπρόσωπε, εσείς προσωπικά και οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου καταδεικνύεται μεγάλη κατανόηση για τα προβλήματα και τις ανάγκες και όλα, για όλα όσα συσχετίζονται με την ΚΕΠΑ την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Είναι μεγάλη τιμή και το γεγονός ότι από πλευρά του Συμβουλίου έχει συνειδητοποιηθεί ότι στην Επιτροπή Εξωτερικών ε, Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνολικά υπάρχει υποστήριξη για τις κοινέ δράσεις ε, και την ε, ανάληψη πρωτοβουλειών από πλευρά των κρατών μελών για την αύξηση της αποτελεσματικότητάς μας στις δράσεις της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, ελπίζω ότι όλοι θα έχουν ακούσει και θα έχουν πληροφορηθεί για αυτά τα οποία είπε ο Ρόμπερτ Γκέιτς, ο Υπουργός ε, ε, Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχε υποστεί επικρίσεις αρχικά. Στη συνέχεια καταδείχθηκε ότι πολλοί Ευρωπαίοι πολιτικοί και πολλοί αξιωματούχοι από πλευράς της Ευρώπης αποφάσισαν δυστυχώς ότι ήταν ε, από πλευράς του η αντιμετώπιση αυτή, η αντιμετώπιση των προκλήσεων, τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά λοιπόν την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας ε, και σε συνεργασία μεταξύ ΕΕ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα όσον αφορά την επικέντρωση σε συνέργειες ε, και κοινέ δράσεις που θα βελτιστοποιήσει την χρήση των κονδυλίων από πλευράς προϋπολογισμού η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση είναι παγκόσμιο φαινόμενο και έτσι έχει επιπτώσεις και στον τομέα της άμυνας που έχει υποστεί συνέπειες. Υπάρχει κοινή τάση για την περικοπή κονδυλίων όσον αφορά κονδυλία για την άμυνα από πλευρά των κρατών μελών και αυτό φυσικά αποτελεί αντικείμενο ανησυχίας για εμάς. Αληθεύει ότι το να διατηρήσουμε τις δράσεις σε σχέση με την άμυνα όταν υπάρχει οικονομική κρίση και όταν υπάρχουν κοινωνικές εντάσεις δεν είναι καθόλου εύκολο εγχείρημα. Αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω, θεωρώ ότι ακόμη και σε τέτοιες ε, ε, περιόδους αναταραχών και κρίσεων δεν θα πρέπει να μελήσουμε, δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε τις ανάγκες τις δημοσιονομικές του τομέα της άμυνας και στην έκθεσή μου αναφέρω κάποιες δυνατότητες να βελτιστοποιήσουμε την χρήση των κονδυλίων ακόμα και αν τα κονδύλια, οι πόροι που έχουμε είναι λιγότεροι από ό,τι σε σχέση με το παρελθόν πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα κονδύλια, αυτούς τους πόρους με τον βέλτιστο τρόπο και αυτό το οποίο είπατε, είπατε οι εκπρόσωπε είναι πολύ σωστό η ιδέα pooling and sharing δηλαδή κοινή συσσόρευση, συνάθρηση προσπαθειών και επιμερισμού έργων, έργου. Αυτό θα βοηθήσει να μειωθούν ε, οι δαπάνε και να ταυτοποιήσουμε και εντοπίσουμε τα ουσιοδέστερα εγχειρήματα από πλευρά στρατηγική μα. Θα πρέπει τελικά να επικεντρωθούμε σε σχέση με τι μεταφορέ, ε, την επιμελητία, λογιστική επιμελητία, ιατρική υποστήριξη και συνδρομή, ε, επιτήρηση και εποπτεία όσον αφορά την χρήση χημικών και βιολογικών όπλων για παράδειγμα, πληροφορίες από πλευράς υπηρεσιών πληροφοριών και κατασκοπίας. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες ε, κοινών προσπαθειών και κοινού επιμερισμού έργου. Δεν μπορούμε να υπερεκτιμήσουμε τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνα ως οργανισμού που θα μπορέσει να δώσει την δυνατότητα να συντονίσουμε καλύτερα τις δράσεις μας ταυτοποιώντας, εντοπίζοντας τις ανάγκες. Και ένα άλλο θέμα όσον αφορά και την τεχνολογική πρόοδο. Υπάρχουν πάλι χωλένουμε πρέπει να πω σε κάποιους τομείς με, σημαντικό, με πολύ έντονο τρόπο. Και όσον αφορά και τις προσφορές ε, για τις ε, συμβάσεις στον τομέα της ε, άμυνας, όλα αυτά τα θέματα προμηθειών και συμβάσεων θα πρέπει να επανεξεταθούν. Μόλις ξεκινήσαμε τη δουλειά και πρέπει να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ. Θα σε ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό στη συνέχεια ο κύριος Τοσενόφσκι παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία, είπατε εκπρόσωπε, εδώ λαμβάνω τον λόγο ως εισηγητής για την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ήτρε για αυτό το θέμα. Είναι πιθανότατο ότι λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης και των συνεπαγόμενων περικοπών των κονδυλίων, τα προγράμματα για την αμυντική βιομηχανία θα υποστούν αρνητικές συνέπειες. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις αυτών των περικοπών μια κοινή αμυντική προσπάθεια έχει νόημα από πλευρά ε, δαπανών. Όμω ε, τίθεται το θέμα κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών. Γι' αυτό η ευρωπαϊκή πολιτική άμυνα πρέπει να οδηγήσει σε μια πολυσχηδή, πολύμορφη συνεργασία, διατηρώντα και διασφαλίζοντα όμω τι εθνικέ ε, ιδιομορφίε και ανάγκε των επιμέρου συμβαλωμένων. Είναι ανάγκη να προβληματιστούμε και να δούμε πώ θα υπάρξει παγίωση τη ζήτηση και αντιμετώπιση με τον βέλτιστο τρόπο τη ζήτηση όσον αφορά κοινέ έρευνε ή την προσπάθεια κάλυψης των αναγκών με κοινό τρόπο. Έχουμε και υπηρεσίε που εξάγουν αλλά άλλε που δεν είναι ικανέ να υποστούν το διεθνή ανταγωνισμό. Αυτέ οι εταιρείε θα πρέπει σε σχέση με την πολυμορφοποίηση του χαρτοφυλακίου του να δράσουν και στην κοινωνία των πολιτών. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τον γύρο αυτών των παρεμβάσεων. Τώρα εξ του ΕΛΚ θα λάβει τον λόγο ο κύριο Μπροκ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, Κυρία Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είπατε εκπρόσωπε συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την προεργασία που έγινε από την δική μας Επιτροπή για την Ασφάλεια και Άμυνα. Είναι σαφές ότι για μας η εξωτερική πολιτική είναι πάντα προληπτικά μέτρα που πρέπει να ε, λαμβάνουμε για τον στρατιωτικό ή αμυντικό τομέα. Αυτή είναι η γραμμή αφετηρίας. Προληπτική δράση για την ειρήνη και την ασφάλεια. Διασφάλιση και διατήρηση της ειρήνης και ασφάλεια. Γι' αυτό είναι αναγκαία η στρατιωτική δράση. Μια και είναι αναγκαία η στρατιωτική δράση πρέπει με τον βέλτιστο τρόπο να χρησιμοποιούνται οι δράσεις μας και να χρησιμοποιούμε τα σωστά μέσα. Η έκθεση καταδεικνύει ότι δεν χρησιμοποιούμε τους πόρους και τα κονδύλια με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Όταν περνάμε μια περίοδο ε, οικονομικής κρίσης και σπανή σπανίδα κονδυλίων πρέπει να δράσουμε αποτελεσματικά. Γι' αυτό για το λευκό βιβλίο που καθορίζει τους στόχους και τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη πλευρά τα κονδύλια τα οποία χρειάζονται για να γίνουν αυτές οι δράσεις στον τομέα των αγορών και στην έρευνα θα πρέπει από κοινού να κάνουμε πολλά περισσότερα από ότι καθένας να ε, εκπονεί τη δική του, τις δικές του σφαίρες ή πυρομαχικά ή εξοπλισμό με ξεχωριστό τρόπο. Από κοινού πρέπει να δράσουμε. Επίσης στον τομέα της ε, εκμετάλλευσης ε, πολυεθνικών ε, μέσων που έχουμε πρέπει να προχωρήσουμε πιο πολύ και να χρησιμοποιήσουμε την λειτουργικότητα και να δούμε τα προβλήματα που υπάρχουν να επανεξεταστούν ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Πρέπει κοινέ προσπάθειες να κάνουμε για την χρήση και προστασία των στρατιωτών μας. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις όσον αφορά το Αφγανιστάν και για την μη ύπαρξη της πιο σωστής συνεργασίας και που από το Βερολίνο για παράδειγμα όσον αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση την βέλτιστη χρήση των πόρων για την ε, αντιμετώπιση κρίσεων ε, τι τις στρατιωτικές μας δράσεις αυτό είναι αναγκαίο υπέρ της ελευθερίας και ασφάλειας και την προάσπιση των στρατιωτών μας. Και κυρία Αντιπρόεδρε, έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε, ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει πολιτική βούληση, πολιτική συλλογική βούληση, ώστε έτσι να μπορέσουμε σε σχέση με τις πρωτεύουσες μας να κινητοποιηθούμε προς την ορθή πορεία. Ευχαριστώ. Για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, για ένα λεπτό, η κυρία Κοπά παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, λέει διάστον η έκθεση που συζητάμε σήμερα και για την οποία θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή τον κύριο Λίζεκ αφορά το μέλλον του αμυντικού τομέα την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Δύο είναι για μας τα βασικά ζητήματα. Αφενός, να φροντίσουμε να ενισχυθούν συνέργειες και συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αποφύγουμε κατασπατάληση πόρων και αφετέρου να διαφυλάξουμε τις θέσεις εργασίας στον αμυντικό τομέα. Η συγκυρία απαιτεί έναν έξυπνο συντονισμό ώστε να μπουν οι βάσει για την ανάπτυξη μια ανταγωνιστική σε διεθνέ επίπεδο βιομηχανία που θα μπορέσει προοπτικά να δημιουργήσει νέε θέσει εργασία στον τομέα τη άμυνα. δυστυχώ η αναδιάρθρωση των αμυντικών βιομηχανιών είναι αναπόφευκτη. αυτό που πρέπει να φροντίσουμε είναι να γίνει με όσο το δυνατόν λιγότερε συνέπειε για την αποσχόληση σε τελική ανάλυση ευρωπαϊκή αλληλεγγύη εξειδίκευση διαλειτουργικότητα και συμπληρωματικότητα είναι για μας οι κατευθυντήριες γραμμές μιας προοδευτικής πολιτικής στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και μια απάντηση στην κρίση. ευχαριστώ. ευχαριστούμε Κόπα για τους ε, δημοκράτες και φιλελεύθερους για δύο λεπτά η κυρία Νικολάη παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπατή εκπρόσωπε, πιστεύω, θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση για την έκθεση ΛΙΖΕΚ, αυτή η συζήτηση που διεξάγουμε είναι αποφασιστική σημασίας για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Είναι μια πολύ καλή έκθεση που αναλύει πολύ σωστά τα θέματα και προτείνει και λύσεις για προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Και πέρα από όλα αυτά είναι μια έκθεση η οποία αφορά την συνοχή και συνεκτικότητα όσον αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Έχουμε την δυνατότητα την κρίση που αντιμετωπίζουμε να την χρησιμοποιήσουμε ως ευκαιρία υπέρ της αμυντικής βιομηχανίας, υπέρ της άμυνας και ασφάλειας. Δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω βέβαια ότι οι περικοπές κονδυλίων όσον αφορά την πολιτική άμυνα αποτελούν, θα μπορούσαν να είναι κίνδυνος για την ε, κοινή μας πολιτική ασφάλειας και άμυνας τα χάσματα τα οποία είναι ήδη σήμερα μεγάλα μεταξύ των κρατών μελών και των κρατών σε, ε, σχέση με το ΝΑΤΟ, κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ΝΑΤΟ ε, μπορούν να αποδυναμώσουν αυτά τα ε, χάσματα και κενά. Ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας ως οργανισμός θα πρέπει ως δυνατότητα να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης από πλευρά μας για να βελτιωθούμε. Η δυνατότητα ολοκλήρωσης και αποτελεσματικότητας πρέπει να βελτιωθεί για το pooling και sharing, για την κοινή προσπάθεια με μέσα και κοινό επιμερισμό έργου, ώστε να υπάρχει διαλειτουργικότητα δράσεων που θα διασφαλίζεται σε μια κοινή πολιτική άμυνα, σε ένα κοινό μηχανισμό άμυνα, με ένα αποτελεσματικότερο τρόπο, διότι υπάρχει ανάγκη παντού παγκόσμια αποστολέ αποστολές από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο στρατιωτικό επίπεδο και στο επίπεδο ασφάλειας. Πρέπει στην Ευρώπη να βελτιώσουμε, να ενισχύσουμε το ερευνητικό δυναμικό σε κάποια κράτη-μέλη και πρέπει περαιτέρω να προσπαθήσουμε και να μεριμνήσουμε, να φροντίσουμε ότι θα έχουμε ένα διαφανές πλαίσιο όσον αφορά τις προμήθειες ε, και ε, την, ε, τις αγορές διότι ένας ευάλωτος, πολύ ευαίσθητος τομέας είναι αυτός επειδή υπάρχει μεγάλο, μεγάλο ποσοστό διαφθοράς υπάρχει ένας διοντολογικός κώδικας για να βελτιωθούν τα πράγματα πρέπει όμως αποτελεσματικά να εφαρμόζεται για να έχουμε τα σωστά αποτελέσματα. Όταν δημιουργείται δυναμικό, πρέπει αυτό το δυναμικό να χρησιμοποιείται προ όφελο των πολιτών και όχι με άλλο τρόπο ει βάρο του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Νικολάη για του πράσινου και την Ευρωπαϊκή Συμμαχία. Ο κύριο Μπουτικόφερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχήν πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Λίζεκ για μια καλή έκθεση. Τον ευχαριστώ λοιπόν που πραγματικά όπως ο Έλμαρ Μπρόκ προανέφερε στην παρέμβασή του, προσπαθεί να δραχθεί της ευκαιρίας που βρίσκεται, που έγκυται στο ότι σε όλους τους εθνικούς προϋπολογισμούς τα κονδύλια είναι μικρότερα, είναι λιγότερα. Και γι' αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί η διασπάθηση κονδυλίων που είχαμε μέχρι σήμερα. Πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Η ευκαιρία της έννοιας pooling και sharing είναι κάτι του οποίου δράτεται ως ευκαιρία ο κύριος Λίσεκ στην έκθεσή του. Και με κάποιες μικρές τροπολογίες προσπαθώ, προσπαθούμε με ιδιαίτερα ευγενικό τρόπο να αυξήσουμε την πίεση έναντι των κρατών μελών για να δράσουμε πιο αποτελεσματικά. Αν γίνουν αυτά τότε θα υπεψηφίσει η ομάδα μου αύριο αυτή την έκθεση. Υπάρχουν όμως δύο θέματα που βρίσκονται στην αρνητική πλευρά αφενός γίνεται η προσπάθεια τώρα δεδομένης ε, της ε, ε πανίδα των κονδυλίων στα κράτη-μέλη να κανιβαλίσουμε τον προϋπολογισμό για την άμυνα, να τον χρησιμοποιήσουμε για άλλους σκοπούς. Δεν είναι σκόπιμο τώρα σε σχέση με στρατιωτικές δαπάνες ε, ή στο πλαίσιο των ε, FP7 του 7ου πλαισίου έρευνας ε, και ανάπτυξης να χρηματοδοτήσουμε δράσεις από αυτά τα κονδύλια. Δεν είναι σωστό να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια αυτά για άλλους σκοπούς ε, ή να χρησιμοποιηθεί από τον προϋπολογισμό μας ένας ε, στρατιωτικός έρασμος ως πρόγραμμα. Πρέπει να μεριμνήσουμε λοιπόν με αποτελεσματικό τρόπο η περικοπή κονδυλίων να αποτελέσει αντικείμενο βέλτιστης απόδοσης και επίδοσης. Και τρίτον, επειδή εδώ έχουμε κάποιες προτάσεις από πλευράς φιλελευθέρων που κατά τα άλλα πάντα είναι υπέρ του ανταγωνισμού, μέσα από αυτή την έκθεση καταβάλλεται με άλλα λόγια η προσπάθεια, τα κεκτημένα τα οποία έχουμε επιτύχει μέσα στο Defense Package, την δέσμη μέτρων για την άμυνα, όσον αφορά την διαφάνεια, όσον αφορά την προκήρυξη προσφορών και ε, διαγωνισμούς, να πάψει να υπάρχει αυτή η διαφάνεια λένε πρέπει να διασφαλίσουμε θέσεις απασχόλησης και με αυτό τον ελιγμό προσπαθούν να ευδοκιμήσει η προσπάθειά τους. Παρακαλώ να μην ενδώσουμε. Έχουμε τροπολογίες που ζητούμε επιμέρους ψήφιση ξεχωριστά παραγράφων. Αυτά τα στοιχεία, αυτές οι προτάσεις δεν πρέπει, δεν πρέπει να ενταχθούν σε αυτή την έκθεση. Αποτελούν συντηρητικά στοιχεία, είναι αναποτελεσματικά και συνεχίζουν την διασπάθηση κονδυλίων. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπιουτικόφερ για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές για δύο λεπτά. Ο κύριος Φανόρντεν παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριο Λίζεκ έχει ετοιμάσει μια λεπτομερέστατη και καλογραμμένη, καλοσταγμένη έκθεση. Δυστυχώ όμω καταλήγει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Φαίνεται ότι κάθε πρόβλημα σε αυτό το σώμα, Πρόεδρε, απαντάτε με την ε, ίδια λογική. Περισσότερη Ευρώπη. Όχι, εδώ θέλουμε περισσότερε θετικέ δυνατότητε και την επίδειξη αλληλεγγύη με τον ΝΑΤΟ για να έχουμε σοβαρέ επιχειρησιακέ δεσμεύσει και την πολιτική βούληση. Αλλά εδώ δεν λείπουν. Αυτά είναι δύο στοιχεία που λείπουν ήδη σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε. δούμε ότι η πραγματική απειλή και οι προκλήσει που έχουμε να αντιμετωπίσουμε δεν θα επιληθούν αν χρησιμοποιήσουμε τι ίδιε διαδικασίε όπω όλα τα άλλα ζητήματα, όπω το ευρώ, και στην άμυνα. Θα πρέπει την ε, πολιτική άμυνα και ασφάλειε να μην ε, παρασυρθούμε τι φιλοδοξίε μα και καταστρέψουμε όσα ήδη έχουμε καταφέρει. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για το κατά πόσον η πολιτική άμυνα και ασφάλεια μπορεί να είναι άστοχη ή όχι και κατά πόσο πρέπει να έρχεται στην ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Ε, κατά πόσον θα πρέπει εδώ να υπάρξει ανάληψη ευθυνών από το ΝΑΤΟ ή όχι. Η περίπτωση τη Λιβύη έδειξε πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι η έννοια αυτή του pooling and sharing, τη εκμετάλλευση και επιμερισμού ικανοτήτων. Τι ε, ευθύνε έχουν οι πολιτικοί ηθήνοντε. Πρόεδρε, φαίνεται ότι από το επιτελείο που εργάστηκε για τη Λιβύη και από τις 28 χώρες που συμφώνησαν στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στη Λιβύη ότι τελικά λιγότερο από το ίμιση συμμετείχαν στην πράξη και λιγότερο από το 1 τρίτο ήταν έτοιμες να πάρουν μέρος σε επιχειρήσεις άμεσης δράσης. Πώς χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Γαλλία να ενισχύσουν άλλους και να παράσχουν ζωτικές στρατιωτικές δυνατότητες. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι με η έκθεση αυτή δείχνει ότι θέλουμε να επιβάλλουμε μια στρατηγική οικονομίας και στην ευρωπαϊκή άμυνα. Ενώ υπάρχουν δυνατότητες ε, στρατιωτικές, υπάρχει δυναμικό, υπάρχει περιθώριο διαλειτουργικότητας και βεβαίως συνεργασίες με τον στρατηγικό μας εταίρο της ΗΠΑ. Σας ευχαριστούμε κύριε Φανόρντεν. Ο κύριος Μπιουτικόφερ σήκωσε μια μπλε κάρτα. Την δέχεστε αυτή την ερώτηση από τον κύριο Μπιουτικόφερ και Φανόρντεν. Δέχεστε. Εντάξει. Προχωρήστε κύριε Μπιουτικόφε στην ερώτησή σας. Αν είσαστε τόσο στεναρά κατά της έννοιας της pooling and sharing που πρότεινα, πώς θα καταφέρετε να συμβιβάσετε το ότι στο ΝΑΤΟ Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει. Η ίδια έννοια εξορθολογισμού προσπαθειών δυναμικού και μέσων. Μόνο υπό διαφορετική έννοια, υπό άλλο τίτλο. Ευχαριστώ. Uh, Mr. Κύριε Μπουτικόφερ, μπορώ να σα προβάλλω και επισήμω το επιχείρημα. Ούτω ή άλλω όλα στο ΝΑΤΟ απειλούνται. Γιατί προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ευθύνε, γιατί προσπαθεί να, να επαναλάβει όσα γίνονται στο ΝΑΤΟ. Είναι απλή επανάληψη όλα αυτά. Ενώ στην ουσία στο ΝΑΤΟ προσφεύγουμε όλοι. Εδώ το μεγάλο πλεονέκτημα του ΝΑΤΟ είναι ότι η διακυβερνητική συμμαχία και τα κυρίαρχα έθνη μπορούν να αποφασίσουν να τα συμμετάσχουν ή όχι σε συγκεκριμένε επιχειρήσει. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα. Και αυτή είναι μεγάλη διαφορά. Τώρα, για το pooling and sharing, το, τη συνεκμετάλλευση και περιορισμό ικανοτήτων. Έχουμε πολλούς συνδυασμού με τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟΥ. Υπάρχει βεβαίω περιθώριο για τη συγκέντρωση και του περιορισμού ικανοτήτων, αλλά σκεφτείτε τι έγινε με το AWACS και την κρίση στη Λιβύη. Εδώ αυτό που χρειαζόμαστε είναι αξιόπιστη στεναρή ε, σύμμαχη που όταν θα τους χρειαστούμε θα εμφανιστούν ακόμη και αν υπάρχουν πολιτικές δυσκολίες και επίσης θα μας παράσχουν τις δυνατότητες ε, για την διεξαγωγή πολέμου και θα ε, μας υποστηρίξουν. Σας ευχαριστούμε κύριε Φανόρντεν για την Ενωτική Ευρωπαϊκή Αριστερά και την Πράσινη Βόρεια Αριστερά για 1,5 λεπτό η κυρία Λούισεν παρακαλώ. Vielen Dank. Σα ευχαριστώ πολύ. Η σημερινή συζήτηση διεξάγεται με παρασκήνιο την χρηματοοικονομική δημοσιονομική κρίση όπου υπονομεύεται η βάση επιβίωσης ε, των ανθρώπων και τα δικαιώματά τους και η δημοκρατία. Και με το παρασκήνιο ότι παγκόσμια μυριάδες ε, άνθρωποι, κυρίως παιδιά, υποσυτίζονται και λιμοκτονούν. Αν πρέπει κάπου να εξοικονομήσουμε κονδύλια στην Ευρώπη, πρέπει στον αμυντικό τομέα να το κάνουμε αυτό. Άμυνα τι σημαίνει. Άμυνα έναντι εξωτερικών υποθέσεων. Ωραίο είναι να πούμε εντάξει, σε αυτό τον τομέα μπορούμε να έχουμε εξοικονόμηση κονδυλίων. Αν καταλήξουμε όμω στην πριτανεύουσα λογική από πάρα πολύ υψηλό επίπεδο αμυντικών δαπανών, φαίνεται ότι υπό πρόσχημα πίεση των δαπανών μεγαλύτερη προσπάθεια θα γίνει ώστε η αμυντική βιομηχανία να έχει ακόμα μεγαλύτερα κέρδη και δραστηριότητες. Πιστεύω ότι το σενάριο μιας απειλής φουσκώνεται ιδιαίτερα από κάποιους και δεν αληθεύει ότι περικοπές στον τομέα της άμυνας θα οδηγήσουν στην περικοπή και απώλεια θέσεων απασχόλησης. Αυτό δεν αληθεύει. Όμως οι υψηλέ δαπάνες παίρνουν κονδύλια από εκεί που χρειαζόμαστε κονδύλια περισσότερο. Οι προτάσεις του κυρίου Λίσεκ σημαίνουν επίσης και ένα κίνδυνο για τη δημοκρατία με τον μη δημοκρατικά ελεγχόμενο μηχανισμό των Αθηνών ή με την ανάμειξη αστικών και στρατιωτικών στόχων και έργων. Εμείς ε, θα έχουμε την, ε, στην ψήφιση αυτή θα έχουμε τη δική μας δυνατότητα να τοποθετηθούμε για το αίτημα ριζοσπαστικού αφοπλισμού και ανάπτυξης του πολιτικού σκέλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Θα ευχαριστούμε κυρία Λόσινγκ για την ε, Συμμαχία υπέρ της Δημοκρατίας για ένα λεπτό. Ο κύριος Τέρον παρακαλώ. Arvoisa puhemies. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πάρα πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε λόγω τη κρίσης βρίσκονται σήμερα στην κατάσταση οι δαπάνες τους να περικόπτονται. Το έκανε και η Φινλανδία, η χώρα μου αυτό. Περιέκοψε δαπάνες και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Η ασφάλεια όμως των πολιτών μας πρέπει να διασφαλίζεται. Δεν μπορεί άλλο έργο να, είναι, να έχει υψηλότερη προτεραιότητα από αυτό. Είναι ανήθικο να υπάρχουν περικοπές στην ασφάλεια όταν δισεκατομμύρια ευρώ ταυτόχρονα δαπανώνται και διασπαθίζονται αλλού για άλλες χρήσεις. Οι περικοπές στον τομέα του προϋπολογισμού της ε, Άμυνας μειώνει επίσης και τη σπουδαιότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια κλίμακα. Για παράδειγμα, σε σχέση με την Αραβική Άνοιξη το είδαμε ότι χρειαζόμαστε και στρατιωτικές παρεμβάσεις, οι ε, στρατιωτικές επεμβάσεις. Η κοινή συνεργασία είναι καλή υπόθεση, αλλά και τα κράτη-μέλη, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαρκώς θα πρέπει να υπενθυμίζουμε ότι αυτή τη συνεργασία πρέπει να την βελτιώσουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για τους μη εγγεγραμμένους θα λάβει τώρα τον λόγο για 1,5 λεπτό ο κύριος Λεπέν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, μπορεί εδώ να ευνηδιάσουμε τους πλέον ομοσπονδιακούς και φεντερλιστές ε, εξημών, όμως ε, η λύση στην πολιτική άμυνας και ασφάλειας είναι εθνική. Τώρα να ψάχνουμε διπλωματική απάντηση σε τέτοια διζητήματα αρμόζει και προσήκει στα έθνη. Εδώ λοιπόν όλα αυτά είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας. Η κοινή διαχείριση στρατιωτικών μέσων είναι μια τεράστια πλάκα. Και τα κράτη-μέλη που πιστεύουν ότι η άμυνά τους μπορεί να σχεδιαστεί στην Ουάσιγκτον σημαίνει ότι ουσιαστικά θα έχουν αμερικανικού εξοπλισμού στα χέρια του. Η Ευρώπη μπορεί να πρικοδοτηθεί και να εφοδιαστεί με τα απαραίτητα σε αυτόν τον τομέα όπω ε, και σε άλλου. Αλλά όχι χάρη στον κοινοτικό προπολογισμό και μόνο. Ούτω ή άλλω, εδώ τίποτε δεν μπορεί να επιληθεί ε, χωρί την διακυβερνητική συνεργασία, όπω έχουμε δει και σε άλλε περιπτώσει. Αλλά δεν φτάνει και δεν χρειάζεται εδώ η αποκλειστική παρέμβαση των Βρυξελών. Λυπάμαι, κυρία Άρθον, αλλά νομίζω αυτό που λέτε είναι σαν αυτό που λέει ο οργανισμός Standard Poor's ε, για την ε, ε, πολιτική της, και για την κατάσταση της οικονομίας μας στους 27 λαούς μπορεί το ζεύγος ε, Μέρκε Σαρκοζή να επιβάλλει αποφάσεις ε, κοινέ. Ας θυμηθούμε τι γινόταν στην Σοβιετική Ένωση ότι σε περιπτώσεις περικοπών δημοσιονομικών η πολιτική άμυνας και πρώτη θυσιάζεται. Ε, και εδώ είναι απερχιωμένα τα συστήματά μας και οι εξοπλισμοί μας πολλές φορές. Λόγω των κλειδονισμών λοιπόν στο χρηματοπιστωτικό ε, σύστημά μας θα πρέπει να δούμε τι κάνουν οι Αμερικάνοι ε, απέναντί μα. Και ο καθένα να αναλάβει τι δικέ του ευθύνε και να καταβάλει τι θυσίε που μπορεί να φέρει ει πέρα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να εξεύρουμε τα αναγκαία μέσα, όχι μόνο για την ασφάλεια και την εθνική άμυνα, αλλά και για τη συνεργασία των μέσων μεταξύ μα για να αντιμετωπίσουμε κοινέ προκλήσει. Να καλύψουμε αδυναμίε και κενά. Αλλά όχι ε, με μπαλώματα, γιατί αυτό ποτέ δεν μα οδήγησε πουθενά. Η... Μπλε κάρτα δείχνετε. Γιατί δεν είναι μπλε αυτό. No. Όχι. Δεν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση στον κύριο Λεπέν. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Θα περάσουμε ένα ειρηνικό, ένα ήρεμο απόγευμα από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, περνάμε σε λοιπούς, στους λοιπούς εγγεγραμμένους ομιλητές. Για δύο λεπτά τώρα έχει το λόγο ο κύριος Ντανζόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η εξαιρετική έκθεση του συναδέλφου Λίζεκ νομίζω ότι μας δείχνει ε, ποιος είναι ο βασικός περιορισμός που βαρύνει ε, τους εθνικούς και πολυμερείς ε, αμυντικούς προπολογισμού, τα δημοσιονομικά προβλήματα δηλαδή που υπάρχουν, αλλά και ένα στρατηγικό σημαντικό στοιχείο είναι η στάση των Αμερικανών φίλων και συμμάχων, οι οποίοι ούτε μπορούν ούτε θέλουν να κάνουν πλέον τα πάντα στη δική μας θέση σε ό,τι αφορά ε, την ασφάλεια, όπως έδειξε πολύ ξεκάθαρη περίπτωση της Λιβύης. Με αυτούς τους περιορισμούς λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να δώσουμε νέα πνοή ε, ε και φιλοδοξία ε, στην κοινή πολιτική άμυνα και ασφάλεια και στο επιχειρησιακό και σε ό,τι αφορά τι δυνατότητες. Για το επιχειρησιακό, είπατε εκπρόσωπος μίλησε γι' αυτό το comprehensive approach και δικαιολογημένα ε, θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε τις ε, διεθνείς κρίσεις, αλλά θα πρέπει και είναι ο ρόλος σας αυτός, αυτή η προσέγγιση να μην ε, θυσιάσει τα στοιχεία της ασφάλειας και ενδεχομένως τα στρατιωτικά. Ε, θα πρέπει να είναι πραγματικά δηλαδή γενική, συνολική αυτή η προσέγγιση και να μην ε, παραγνωρίζει το στοιχείο της ασφάλειας. Όπως είπατε για το κέρας της Αφρικής και το Σαχέλ που αν κατάλαβα καλά λέτε να γίνουν εκεί αποστολές. Τώρα θα πρέπει να χαιρετήσουμε τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Υπάρχουν βέβαια κάποιες εμπλοκές και προβλήματα με τον προπολογισμό. Σας ευχαριστούμε και σας παρακαλούμε να μας ε, μεταφέρετε τις εκτιμήσεις σας για τις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Και να πω ότι σε ό,τι αφορά την αμυντική βιομηχανία η ενοποίηση, η παγίωση, η ενίσχυση των ε, ημαντικών ε, αμυντικών βιομηχανιών, αλλά και ο εξορθολογισμός τους θα συνεπάγεται και τη στήριξη της απασχόλησης αλλά και των τεχνολογιών που υπερβαίνουν τον τομέα αυτό. Είναι στρατηγική σημασία για τις οικονομίες μας γενικότερα, ιδίω εν καιρό κρίσης. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντανζόν. Για ένα λεπτό έχει το λόγο ο κύριος Γκουαλτιέρη τώρα. Ευχαριστώ το είπε η κυρία Κοπά. Ε, η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στηρίζει την έκθεση Λίζεκ. Εδώ νομίζω έχουμε ένα μικρό αλλά σημαντικό βήμα πρόοδου. Ε, από τις προτάσεις του Συμβουλίου. Περίμενε περισσότερα βέβαια το Κοινοβούλιο, κυρίως για τις κοινέ δυνατότητες συντονισμένης ε, διεξαγωγής επιχειρήσεων. Αλλά η πραγματική εγκατάλειψη της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας τελικά αποφεύχθηκε. Ευχαριστώ λοιπόν την είπατε εκπρόσωπο για τη δουλειά της σε αυτό το μέτωπο. Μιλάμε εδώ τώρα για επιχειρήσεις. Εάν σκεφτούμε και τι έγινε με την ε, όχι τόσο κατησυχαστική περίπτωση της Λιβύης και τη U4 ή το Σουδάν και το Σαχέλ. Θα πρέπει λοιπόν να αποτιμήσουμε τα αποτελέσματα αυτά και να είμαστε έτοιμοι για πολιτική και δημοσιονομική στήριξη. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία ήδη εφαρμόζονται για τις δυνατότητες συντονισμένου σχεδιασμού και βεβαίω τη ε, αξιοποίηση των ε, στρατιωτικών πόρων. Το Συμβούλιο έχει την βούληση να ενεργοποιήσει κέντρα ε, λήψη αποφάσεων, αλλά μόνο σε μια πρώτη φάση. Δεν θα πρέπει εδώ να χάσουμε την όθηση που ήδη έχουμε, την ορμή και να, μας μα διαφύγουν τα επόμενα στάδια ανάπτυξη. Χρειάζεται λοιπόν εδώ συνολική αποτίμηση. Ευχαριστούμε κύριε Γκουαλτιέρη. Για ένα λεπτό η κυρία Νέιτ Ούτεμπουργκ. Uh, Κυρία Υπάρτη εκπρόσωπε, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή Λίζεκ για την εξαιρετική του έκθεση και να πω κατά δεύτερον ότι ιδιαίτερα εκτίμησα και τα σχόλια που κάνατε εσείς ως απάντηση στην έκθεση αυτή. Έχουμε αυτή την ε, προσέγγιση, pooling and sharing, τη συνεργασία, πώς θα κάνουμε περισσότερα με λιγότερα. Εγώ θα ήθελα ε, να δω πώς ε, θα μπορούσαμε να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των πυρηνικών όπλων. Όλο αυτό το θέμα το ελέγχου των όπλων και δι των πυρηνικών για να μην μιλήσω για την αποπυρηνικοποίηση, ε, αυτό το θέμα ε, σαν να μην υπάρχει. Δεν το βλέπουμε στα ραντάρ μας, σαν εξαφανίστηκε. Πρέπει λοιπόν να, βιωθούν, να αναβιωθούν οι προσπάθειες συγγνώμη, στον τομέα αυτό. Εκεί θα ήθελα να εμβαθύνω εγώ. Μιλάμε για, την, ε, για, τον πυρηνικό αφοπλισμό στη Μέση Ανατολή. Θα είναι Χριστούγεννα όπου να είναι. Ίσως αυτό θα έπρεπε να είναι η ευχή μας για τα Χριστούγεννα. Ένας κόσμος χωρίς πυρηνικά. Ευχαριστούμε την κυρία Νέιτς. Τώρα για ένα λεπτό η κυρία Τζαβέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέει διάστον, Η πατρίδα μου η Ελλάδα οφείλει το 1 πέμπτο του χρέους της στις αμυντικές βιομηχανίες. Όπως ξέρετε υπάρχει το κάζους μπέλι της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδος και οφείλουμε να είμαστε αμυντικά εξοπλισμένοι. Λέει διάστον, δεν μπορούμε πλέον να διατηρήσουμε αυτή την αμυντική πλευρά που είχαμε. Και σας θέτω ένα ερώτημα. Σε περίπτωση που υλοποιεί το κάζους Μπέιλι η Τουρκία, όπως έκανε στο πρόσφατο παρελθόν, ποιος θα μηνθεί των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ μιλάμε για μια πραγματική απειλή, για την οποία χρειαζόμαστε να έχουμε μια αξιόμαχη άμυνα. Θα θέλαμε, λέει Διάστον, αυτό το ποσό και αυτό το προϋπολογισμό να τον αναλάβει η Επιτροπή όταν μιλάμε για μια πραγματική απειλή και όχι για θέμα γοήτρου αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμμετάσχει στο Αφγανιστάν ή εδώ ή εκεί. Υπάρχει μια πραγματική απειλή στην οποία δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε και θα έπρεπε να σκεφτείτε πώς θα ανταποκριθούμε ως Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ε, ο κύριος Βανόρντεν θέλει κυρία Τζαβέλα να σας θέσει μια ερώτηση. Κύριε Βανόρντεν, 30 δευτερόλεπτα έχετε στη διάθεσή σας κύριε Βανόρντεν. Απλά λίγο ναι. ε, περδεύτηκα. Θα μπορούσατε ίσως να μου διευκρινίσετε αυτό που είπατε. Φυσικά και υπάρχουν πραγματικές απειλές και φυσικά πρέπει να έχουμε την κατάλληλη άμυνα. Αλλά ε, το ΝΑΤΟ δεν την παρέχει αυτή την ε, άμυνα. Ε, τελικά τι προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια σχέση. Αυτό που πάει να κάνει δεν σχετίζεται με αυτό που λέτε. Δεν νομίζω ότι για πολιτικά περίεργη και στρατιωτικά ανίκανη οργάνωση δεν νομίζω ότι είπα θα, θα το προτιμούσαν αυτό. Μιλάμε για κοινή ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας. Σε αυτό αναφέρομαι, η οποία είναι ανύπαρκτη όσον αφορά την πατρίδα μου την Ελλάδα, που είναι 30 χρόνια τώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν υπήρξε στρατιωτικό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας πριν από μερικά χρόνια, δεν ήταν το ΝΑΤΟ, δεν ήταν η ευρωπαϊκή ένωση η οποία ανταποκρίθηκε και βοήθησε ήταν ο έκτος αμερικανικός στόλος και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. ελπίζω να απάντησα στην ερώτησή σας κύριε van και μιλάω για υπαρκτό κίνδυνο και όχι για όλα αυτά τα οποία μιλήσαμε εδώ ευτυχώς και αναφέρονται μόνο σε θέματα γοήτρου. ευτυχώς που όλοι εσείς οι άλλοι δεν έχετε το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε εμείς. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό η κυρία Ντότς παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Κυρία είπατε εκπρόσωπε. Εγώ αυτό το απόγευμα θα απόσχω στο να επικεντρωθώ στην ανάγκη σύνεσης ε, και νυφαλιότητα σε δύσκολες περιόδους χρηματοοικονομικές και για την υποστήριξη του ΝΑΤΟ περισσότερο με απλά λόγια και όχι με την περίπλοκη διατύπωση του κυρίου Φανόρντεν. Αλλά κυρία είπατε εκπρόσωπε, εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ένα πολύ ξεχωριστό εξειδικευμένο σημείο το οποίο αναφέρατε στις εισαγωγικέ παρατηρήσεις σας. Την προσυπογραφή του πλαισίου με τη ΣΥΠΑ για τις πολιτικές αποστολές στο Κωσικοπέδιο και Αφγανιστάν και έναν αριθμό ατόμων που εργάζονται σε αυτά τα προγράμματα δραστήρια από τη ΣΥΠΑ. Όλοι πρέπει να καλοχαιρετήσουμε την πραγματογνωμοσύνη αυτών των ανθρώπων από τη ΣΥΠΑ και το θάρρος τους, τη γενναιότητά του σε δύσκολες περιόδους. Ιδιαίτερα η ειδική συγκυρία όσον αφορά την ε, ε, αστυνομία, την ε, αστυνομία από την Βόρεια Ιρλανδία και στο Ιράκ και την εκπαίδευση των αστυνομικών δυνάμεων εκεί και την κατάρτιση των πολιτών ώστε να διασφαλιστεί η ειρήνη και η ασφάλεια μετά την αποχώρηση των Βρετανικών και Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από αυτή τη χώρα. Και βλέπουμε ιδιαίτερα σε μια πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη δουλειά και ιδιαίτερα που δυσχεραίνεται και καθίσταται πιο περίπλοκη από την γραφειοκρατία της Ευρώπης, τη γραφειοκρατία από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα εκείνοι που υπηρετούν στο Αφγανιστάν και το Κωσυφοπαίδιο να μην παρακολύονται με τον ίδιο τρόπο από τους γραφειοκράτες των Βρυξελών. Ευχαριστώ. Θα σε ευχαριστούμε κυρία Ντότς. Θα λάβει τώρα τον λόγο για δύο λεπτά ο κύριος Γκάλερ παρακαλώ. Ναι σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ καταρχήν να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Λίσεκ για την πραγματικά εξαιρετική του έκθεση που θέτει τον δάκτυλο επί του τύπου των ύλων, εκεί όπου υπάρχουν ελλείψεις και κενά και καταδεικνύει πώς και πού μπορούμε καλύτερα να είμαστε πιο αποτελεσματικοί από κοινού. Σωστά αναφέρθηκε ότι η ΚΕΠΑ, η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, μπορεί να είναι μόνο τόσο καλή όσο επιτρέπουμε. Σωστό αυτό ως θέση. Θα έλπιζα ότι την 1η Δεκεμβρίου στα συμπεράσματα του Συμβουλίου περισσότερα θα μπορούσαμε να είχαμε πει και να είχαμε εγκρίνει για παράδειγμα στον τομέα του σχεδιασμού και της αποδοτικότητας καταφέραμε μόλις και μόνο να συμφωνήσουμε ότι το επιτελείο θα ε, βρίσκεται στις Βρυξέλλες αυτό όλο και όλο και όχι, το, όχι συστηματικά ή μόνιμα, αυτό είναι κάτι θλιβερό πρέπει να πω. Δεν καταφέραμε πιο πολλά. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, ναι μεν τοποθετούνται για τα battle groups, αλλά είναι ανήμπορα τα κράτη-μέλη ε, σε σχέση με την περίοδο πριν από το 2012 να διασφαλίσουν κάτι πάνω από δύο battle groups. Σε τι οφείλεται αυτό. Και η πρωτοβουλία pooling και sharing επανειλημμένα αναφέρθηκε αυτή. Την θεωρώ εξαιρετική πρέπει να πω και όχι μόνο υποτασσόμενοι στις ανάγκες ε, και ε, καθήκοντά μας αλλά επειδή πραγματικά μας βοηθά να ενωθούμε και να συγκλίνουμε περισσότερο. Αλλά διαρωτώ η πρωτοβουλία της Γκέντ, της Γάνδης και η πρωτοβουλία pooling και sharing κατά πόσον έχει βοηθήσει τα κενά και χάσματα που υπάρχουν όσον αφορά τα όσα είχαμε διαπιστώσει το 2010 να καλυφθούν να πληρωθούν. Και διαρωτώ με πότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο η δομημένη, διαρθρωμένη συνεργασία θα ξεκινήσει να λειτουργεί. Τι θα γίνει σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2011, αυτά τα οποία είχαμε ζητήσει να γίνουν. Ποια διαβήματα και βήματα ε, διενεργεί και κάνει η εξωτερική υπηρεσία ώστε να υποστηρίξει αυτή τη συνιστόσα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Γκάλερ. Τώρα θα λάβει τον λόγο για ένα λεπτό ο κύριος Πάσκου, παρακαλώ. Η σημερινή προσπάθεια να σώσουμε το ευρώ έχει επιπτώσεις και στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας και αυτά πρέπει να τα προσέξουμε. Πρώτα απ' όλα σκεφτήκαμε την ε, πειθαρχία τη δημοσιονομική η οποία βεβαίως πιέζει τους εθνικούς μας προϋπολογισμούς ενώ συσσωρεύονται οι στρατιωτικές προκλήσεις και μάλιστα στην άμεση και την κοντινή γειτονιά μας. Εδώ λοιπόν υπάρχουν άμεσες απειλές αλλά αντιμετωπίζουμε και ενδεχόμενο συνδυασμό των κινδύνων στο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να σκεφτεί την περιουσιακά στοιχεία διαθέτηση στον δικό τομέα και γιατί πολλοί σε μη φιλικού ε, αγοραστέ. Θα πρέπει να, φτάνουν, να μην φτάνουν οι ευρωπαϊκοί εξοπλισμοί σε λάθο χέρια. Βεβαίω, οι προσπάθειε να σωθεί η Ευρωζώνη έχει ήδη υπονομεύσει την εσωτερική αλληλεγγύη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται λίγοι να συγκεντρώνουν την εξουσία στα χέρια των χωρών τη Ευρωζώνη κυρίω και αυτό ενδεχομένω δεν θα ευνοήσει τι προσπάθειε τη ε, συγκέντρωση και του επιμερισμού ικανοτήτων. Έπειτα, οι Ηνωμένε Πολιτείε μειώνουν την την ε, ε, συνεισφορά του στο ΝΑΤΟ και μιλούν για μια περιορισμένη συμμαχία, όπω ήδη συζητιέται στι δύο πλευρέ του Ατλαντικού. Θα χάσουν όμω έτσι ένα μεγάλο μέρο τη ε, στήριξή του οι ευρωπαϊκέ χώρε. Σα ευχαριστούμε κύριε Πάσκου. Τώρα θα λάβει τον λόγο για ένα λεπτό κύριο Λάμστορφ, παρακαλώ. Ναι, προτού όμω εδώ τοποθετηθώ για αυτό το θέμα, θέλω την παρουσία του πρώην συναδέλφου και αντιπροέδρου Σταύρου Λαμπρινίδη να την επισημάνω και Τώρα δεν ε, μας παρακολουθεί, και δεν καταλαβαίνει βέβαια γερμανικά, δεν φορέ τα ε, ακουστικά. Όταν έχω μια εκδήλωση στο, στον κύκλο ψηφοφόρων μου, στον εκλογικό μου κύκλο, ερωτώ, ερω, γίνεται, υποβάλλεται η ερώτηση ποιο έχει πιο πολλού στρατιώτε, η ΕΠΑ ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απάντηση είναι σταθερά λανθασμένη. Τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν 2 εκατομμύρια στρατιώτε, οι Αμερικανοί 1,4 εκατομμύρια στρατιώτε. Είμαστε οπλισμένοι μέχρι τα δόντια. Όμω ε, σε σχέση με τι δαπάνε μα έχουμε τεράστια ε, βάρη. Το pooling sharing είναι λογική υπόθεση. Δεν μπορούμε όμως να αφήσουμε αυτή την υπόθεση αποκλειστικά στους στρατιωτικούς. Πρέπει πολιτικά να παρακολουθήσουμε τα πράγματα. Γι' αυτό αυτή η έκθεση είναι μεγάλη συνεισφορά ε, υπέρ της πολιτικής συζήτησης και ρύθμισης των πραγμάτων. Ευχαριστούμε τον κύριο Λίσεκ. Θα ήθελα να πω ότι η τοποθέτηση μπορεί το νομικά δεσμευτικό για μια κατεύθυνση όσον αφορά τις προμήθειες και αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις προτεραιότητες. Είναι αποφασιστικό να τηρήσουμε αυτές τις, ανα... Ε, διαδικασίες. Είτε είναι στρατιωτικές είτε αφορούν ε, τον ε, αστικό τομέα υπάρχει η δυνατότητα στρεβλώσεων και γι' αυτό είναι σημαντικό να τονίσουμε αυτή την πτυχή, να παραμείνουμε και να ψηφίσουμε να ρυθμίσουμε αυτό το θέμα έτσι. Ευχαριστώ. Μια στιγμή κύριε Κάρα γιατί ο κύριος Φανόρντεν σήκωσε την μπλε κάρτα θέλει να παρέμβει. Κύριε Φανόρντεν, έχετε μισό λεπτό στη διάθεσή σα. Πρόεδρε, είναι για ενημέρωση η παρέμβασή μου, για πληροφόρηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει στρατιώτε, εντάξει, δεν έχει στρατιώτε στη διάθεσή της. Κανέναν ένοπλο. Απολύτως. Υπάρχουν στρατιώτε στις ένοπλες δυνάμεις των κρατών μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει στρατό. Να, να είναι απόλυτα σαφέ αυτό. Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε λοιπόν την... Αν προσπαθήσουμε έτσι να κάνουμε τη σύγκριση με τη ΣΥΠΑ, δεν λειτουργεί η αναλογία. Ο κύριος ε, Λάμστοφ, μια και ξέρω την ποιότητα των διερμηνέων μας και είναι εξαιρετική, δεν φταίει η διερμηνία. Πρέπει ε, θέμα κατανόησης να είναι αγαπητέ Τζόφρι Φανόρντεν. Είπα, τα κράτη-μέλη έχουν ε, αυτά τα εκατομμύρια στρατιώτες ε, και σε σχέση με τις αμερικανικές δαπάνες δεν έχει νόημα να διατηρηθεί μια τέτοια κατάσταση. Και το pooling και sharing σε σχέση με τους Γάλλους για παράδειγμα, στη στρατηγική πλατφόρμα για τις πυρηνικές δοκιμές όσον αφορά τα αεροπλανοφόρα. Η συζήτηση είναι πάρα πολύ σημαντική και ευχαριστώ τον κύριο Λίσεκ για την πολύ καλή του έκθεση. Για 1,5 λεπτό τώρα ο κύριος Κάρας παρακαλώ. Ναι κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν τρία γεγονότα αδιαμφισβήτητα. Πρώτο γεγονός, η Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε ως εγχείρημα και πρωτοβουλία υπέρ της ειρήνης ώστε να μην γίνονται πλέον στο μέλλον πολεμικές αντιπαραθέσεις και πόλεμοι μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το στόχο, σε αυτό το στόχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 100% τον επιτελέσαμε, τον υλοποιήσαμε. Δεύτερο γεγονός. Παρόλα αυτά, σε όλα τα κράτη-μέλη εξακολουθούμε να έχουμε αμυντικές δυνάμεις και αμυντική πολιτική από πλευρά των κρατών μας. Όπου σε όλα τα κράτη μεταξύ τριών σημείων έχουμε ένα πρόβλημα αποτελεσματικότητας, ένα πρόβλημα στελέχωσης και προσλήψεων και έχουμε και πρόβλημα χρηματοδότησης. Τρίτο επιπλέον γεγονός. Δεν υπάρχει κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνα. Τουλάχιστον δεν υπάρχει αποτελεσματική και πα, αξιόπιστη. χωρίς να υπάρχει μια κοινή πολιτική για την άμυνα και τι ε, αμυντικές δαπάνες και στρατιωτικά όλα πρέπει με βάση αυτά τα γεγονότα να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να υπάρξει αυτή η, άμυν, η κοινή κοινοτική πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Και δείχνει τη σωστή πορεία η έκθεση Λίσεκ ότι μπορούμε όλα να τα κάνουμε σωστά με βάση τις σημερινές υφιστάμενες συνθήκες να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά μας να ενισχυθεί η πολιτική μας αξιοπιστία και δημοσιονομικά οι δαπάνες να μειωθούν όσον αφορά τα κονδύλια. Επειδή από κοινού με τις προσπάθειές μας θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί από ό,τι καθένας από εμάς χωριστά. Ευχαριστώ. Θα σε ευχαριστούμε κύριε Κάρας. Τώρα στη συνέχεια για ένα λεπτό η κυρία Γκόμες παρακαλώ. Οβερμάιερ, hm? έχετε τον λόγο κύριε Οβερμάιερ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Για αυτό το θέμα προφανώς ε, οι μπλε κάρτες που ε, ζητήθηκαν. Θέλω να ζητήσω από τον κύριο Κάρας να δώσει μια απάντηση. Σωστά αναφέρθηκε σε μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας που δεν είναι αποτελεσματική Μπορούμε να το δεχτούμε αυτό αν θέλουμε. Όμως αυτά που αφορούν στην ανάλυση του είδαμε να απουσιάζει ένα στοιχείο στη σωστή τοποθέτηση. Κύριε Κάρας, τι προτείνετε. Μια κοινή πολιτική άμυνας να έχουμε στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τι προτείνετε. Όλα τα κράτη το ΝΑΤΟ εκεί να ε, επικαλύπτουν, να καλύπτουν τις ανάγκες τους και ως εταίροι στο ΝΑΤΟ να δρουν. Ευχαριστώ. Κύριε Κάρας έχετε τον λόγο να απαντήσετε. Μισό λεπτό. Προτείνω πρώτον λέει ο κύριος Κάρας το, περιεχόμενο της έκθεσης ΛΙΣΕΚ να μεταφραστεί σε δράσεις και από εμάς να υποστηριχθεί και να γίνει το νιωστό τμήμα της πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Έχουμε τις συνθήκες Λισαβόνας που ήδη έχουμε δημιουργήσει με αυτήν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας. Πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν σε αυτή την πορεία με άλλες δράσεις. Προτείνω επίσης αυτά τα οποία αναφέρονται να ενισχύσουν τη συνεργασία μας μεταξύ μας. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας, Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση και Ευρωπαϊκή Ένωση Ασφάλειας. Εδώ με βάση τις δυνατότητες των συνθήκων πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να είμαστε συνεπείς. Η έκθεση Λίσεκ δίνει τα σωστά θεμέλια γι' αυτό. Η κυρία Γκόμες τώρα ένα λεπτό παρακαλώ. Η δημοσιονομική κρίση έχει σοβαρές ε, και επικίνδυνες συνέπειες στις δυνατότητες, τις εθνικές, της άμυνας και ασφάλειας και επηρεάζει βεβαίως και την ε, δυνατότητα εκδίπλωσης της ε, κοινή πολιτικής ασφαλείας και άμυνας. Φαίνεται ότι υπάρχει διαρκής πίεση στην αγορά για τους εξοπλισμούς τεχνολογίες ε, τη άμυνα και τη ασφάλεια που αναπτύσσονται στην Ευρώπη. Η πολύ καλή έκθεση του συναδέλφου Λίζεκ τονίζει ότι η συγκέντρωση και επιμερισμό των ικανοτήτων ε, των στατιωτικών εξοπλισμών είναι καθοριστική σημασία για τα ευρωπαϊκά κράτη, ακόμη και εντό του ΝΑΤΟ, όπω κάποιοι παρατήρησαν ασφαλμένα. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ευρωπαϊκή προτίμηση για παρόμοια μέτρα έναντι άλλων. Αλλιώ δεν θα δημιουργηθεί ποτέ η ευρωπαϊκή βιομηχανία που χρειάζεται για να διασφαλίσουμε τη στατική μα ανεξαρτησία και αυτονομία, ώστε να έχουμε μετά σχέσει συνεργασία με άλλου, όπω τον ΟΗΕ, τον ΝΑΤΟ και το καθεξή. Το να υπάρχει διασπάθηση, το να μάλλον υπάρχει δαπάνη ευφυή των συνδετικών πόρων είναι σημαντικό. Και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε ούτε την παράκαμψη, ούτε την αδιαφάνεια του συστήματο. Δεν θα πρέπει να υπάρξει αδυναμία ούτε για να ωφεληθεί η Γαλλία, ούτε για να δημιουργούνται πυρηνικά οπλοστάσια που μπορεί να εξυπηρετούν τα συμφέροντα μεμονωμένων χωρών. Αυτό δεν βοηθά την Ευρώπη να αντιμετωπίσει τι παγκόσμιε προκλήσει προκλήσει που αντιμετωπίζουν. Το αντίθετο. Η Λιβύη, κυρία Άστον, ήταν μια τεράστια χαμένη ευκαιρία για να πετύχει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι η Γαλλο-Βρετανική Συμμαχία. Έπρεπε εδώ να πιστούν τα κράτη-μέλη να μην χάνουν τέτοιε ευκαιρίε, να μην χάνουν τέτοιε δυνατότητε. Εμεί ω Ευρωκοινοβούλιο θα σα στηρίξουμε σε αυτέ τι προσπάθειε. Ευχαριστούμε κυρία Γκόμε. Για 1,5 λεπτό ο κύριο Πρέντα. Σε ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η χρηματοοικονομική, δημοσιονομική κρίση μα κατέδειξε με σαφέστερο τρόπο από ότι οποτεδήποτε στο παρελθόν ότι έχουμε δύο δυνατότητε. Είτε θα διχαστούμε και θα χάσουμε την ολοκλήρωση ή θα μείνουμε ενωμένοι και θα συνεχίσουμε αποτελεσματικά. Η δεύτερη εναλλακτική λύση πιστεύω εγώ ότι είναι η εναλλακτική λύση που θα πρέπει να προτιμήσουμε. Διότι στο τέλο τέλο, σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο πρέπει παγκοσμιοποιημένα, παγκοσμιοποιημένα ενωμένοι να δράσουμε ο προπολογισμό για την άμυνα της Κίνας τα τελευταία χρόνια κατά 200% αυξήθηκε και ταυτόχρονα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις δικές τους αμυντικές δαπάνες ουσιαστικά τις ε, κατέβασαν σε μηδενικό επίπεδο. Χρειαζόμαστε ένα καλύτερο συντονισμό όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλεια. Πρέπει να ενώσουμε το δυναμικό μας και να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες. Η κρίση στη Λιβύη και οι δράση στη Λιβύη κατέδειξαν γιατί πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Καταβάλουμε προσπάθειες στο ΝΑΤΟ. Εντάξει. Χρειαζόμαστε όμως ε, πραγματικά μια αυθεντική δυνατότητα αυθεντικού δυναμικού στην άμυνα. Στην έκθεση συγκεκριμένα βήματα και διαβήματα προτείνονται. Τρία στοιχεία είναι σημαντικά ως άξονες. Καταρχήν ένα ευρωπαϊκό εξάμεινο για την εκπόνηση της πολιτικής άμυνας και ασφάλειας από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, ένας τομέας για την ασφάλεια στο πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης. Και τρίτον, ένα στρατιωτικό πρόγραμμα έρασμος για την, τον καλύτερο καλύτερο σε εισαγωγικά πολιτισμό στα στρατιωτικά και στην άμυνα. Εκφράζω συγχαρητήρια για την εξαιρετική του έκθεση προς τον κύριο Λίσεκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό κύριος Μαφρονικόλας. Μια τέτοια έκθεση είναι απαραίτητη ειδικά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε και συμμεριζόμαστε τους ευρύτερους στόχους της. Τα κράτη-μέλη πρέπει να συνεργαστούν στενότερα και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των κοινών απειλών που εντοπίζονται στην ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας αναλαμβάνοντας το μερίδιο ευθυνών που τους αναλογεί για την εδραίωση της ειρήνης και της ασφάλειας όχι μόνο στην ευρώπη αλλά και στις γειτονικές χώρες και τον ευρύτερο κόσμο η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση μπορούν να αποτελέσουν πρόκληση και συνάμα ευκαιρία για την ολοκλήρωση των αμυντικών πολιτικών της ευρωπαϊκής ένωσης αφού μπορεί να οθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αναγκαίες και σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας. είναι απόλυτα κατανοητό και ενισχύομαι και στηρίζουμε την πολιτική του pooling and sharing για τα σημερινά δεδομένα λόγω όμως της στρατιωτικής κατοχής της κύπρου και της συνεχιζόμενης παρουσίας τουρκικών στρατευμάτων στο νησί η κυπριακή δημοκρατία δεν μπορεί να υλοποιήσει στον βαθμό που θέλει τις εισηγήσεις της έκθεσης ειδικά στον τομέα του pooling and sharing. η κύπρος είναι αναγκασμένη να συνεχίσει να δίδει απόλυτη έμφαση στα δεδομένα με γνώμονα που έχουν το territorial defence την άμυνα δηλαδή της περιοχής. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Συνεχίζουμε με τον κύριο Κέλαμ. Ένα λεπτό και τρία δεύτερα, κύριε Κέλαμ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Γεια σας, κύριε Υπατή εκπρόσωπε. Εξαιρετική έκθεση του συναδέλφου Λίζεκ. Νομίζω καθιστά σαφές ε, το εξής η μείωση του αμυντικού τομέα αποτέλεσμα, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης ουσιαστικά ε, πληγώνει την αξιοπιστία της Ένωσης σαν ε, σταθεροποιητικής δύναμης στον κόσμο. Και δεν είναι μόνο το θέμα της μείωσης των αμυντικών δαπανών. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι οι τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούνται τα κονδύλια δεν υπάρχει συντονισμός ε, στον εθνικό αμυντικό σχεδιασμό και εκεί ε, οφείλονται ε, τα κενά, τα χάσματα ή αλληλεπικαλύψεις. Θα πρέπει να υπάρχει όμως σίγουρα έλεγχος των δαπανών, αλλά αυτό που μας δίνει ως μήνυμα η έκθεση είναι ότι η χρηματοοικονομική κρίση μας δίνει και ευκαιρίες. Είναι καιρός να πάψει η παράδοση του απομονωτισμού, της απομόνωσης ε, στον αμυντικό σχεδιασμό. Και συμφωνώ πλήρω με την υπατή εκπρόσωπο που είπε ότι η πολυεθνική, η πολυκρατική συνεργασία, το pooling και sharing θα πρέπει να είναι κανόνας και όχι εξαίρεση στις δραστηριότητές μας. Θα ήθελα όμως επίσης να μιλήσω για την ε, κυβερνοάμυνα. Είναι ένα τομέα όπου απαιτείται να γίνει κάτι πάρα πολύ ε, ρηξικέλευτο. Πρέπει να έχουμε μοντέρνα σκέψη και αντιμετώπιση της κατάστασης καλή συνεργασία, καλύτερο συντονισμό. Αυτέ είναι οι λέξει κλειδιά και δεν είναι ευσεβισπόθη. Γιατί έχουμε πραγματικά ε, πολύ ζωφερές απειλές ε, επιθέσεων ε, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και θα πρέπει να έχουμε κοινέ ασκήσεις για την αντιμετώπιση επιθέσεων και να αναλύουμε τέτοια σενάρια. Αυτό είναι καθήκον για όλους μας. Και επίσης θέλουμε να υπάρχει ένας Ευρωπαίος συντονιστής για θέματα κυβερνοάμυνας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής, 1,5 λεπτό, ο κύριος Κουμουτσάκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η βαθιά οικονομική κρίση ασκεί πολύ μεγάλες πιέσεις στους εθνικούς αμυντικούς προϋπολογισμούς και κατ' επέκταση στην αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης. Όλοι, ακόμα και τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες και ανελαστικά υψηλέ εθνικές ανάγκες ασφάλεια, όπως η ελλάδα στα ανατολικά της σύνορα αναζητούν ρεαλιστικές και αποτελεσματικές λύσεις στη βάση της λογικής lower cost higher performance. σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες δεν υπάρχουν πολλές επιλογές αυτή είναι η αλήθεια. η μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη αμυντική ευρωπαϊκή συνεργασία είναι έτσι μονόδρομος. είναι όμως ανηφορικός μονόδρομος η εφαρμογή συνεργασίας και συνέργειας δεν είναι απλό εγχείρημα καθώς η αμυντική πολιτική βρίσκεται στο σκληρό πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας των κρατών. γι' αυτό οφείλουμε να εργαστούμε ταυτόχρονα με αποφασιστικότητα αλλά και ευελιξία και γι' αυτό θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη λογική pooling and sharing η οποία γίνεται από επιλογή αναγκαιότητα. ταυτόχρονα βέβαια ειδική σημασία έχουν η διαλειτουργικότητα η συμπληρωματικότητα και βέβαια ο εξορθολογισμός των αμυντικών δαπανών. στην ελλάδα επιχειρούμε να το επιτύχουμε αλλά πιστέψτε με ότι είναι πολύ δύσκολο γιατί αντιμετωπίζουμε υπαρκτή απειλή. με αυτές τις σκέψεις θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο κύριο Λίζεκ για την εξαίρετη έκθεσή του. Ευχαριστώ πολύ σε ευχαριστούμε πολύ κύριε Κουμουτσάκο. Και έτσι ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των αγοριτών και θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία Catch the Eye τώρα πια. Έχουμε ονόματα περισσότερα, περισσότερων ευρωβουλευτών από εκείνους που μπορούν να παρέμβουν. Από κάθε κοινοβουλευτική ομάδα ένας, ο κύριος Κέλλη πρώτος. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο, κύριε Κέρ. Ευχαριστώ. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν θα είχαμε και ανάγκη από στρατιωτικέ δυνάμει. Αυτό θα ήταν το όνειρο του καθενό στον κόσμο μα, αλλά ο κόσμο γίνεται καθημερινά και πιο επικίνδυνο. Οπότε αυτό φαίνεται ότι και στο μέλλον θα συνεχίσει, θα συνεχίσει να ισχύει. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία στην κυκλοφορία των πολιτών, των ανθρώπων, αλλά και περισσότερε ευκαιρίε για του τρομοκράτε και τι οργανώσει του να προβούν σε απόπειρε δολοφονικέ. Εδώ λοιπόν θα πρέπει και εμεί να λάβουμε το ρόλο μα για να υπερασπιστούμε τι θετικέ δυνάμει, να υπερασπιστούμε του πολίτε και να προλάβουμε τι εγκληματικέ οργανώσει και τι συμμορίε ε, των κακοποιών. Εδώ λοιπόν σκεφτείτε ένα απλό παράδειγμα. Τα τσιγάρα που έχουν καταναλωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καθαρεί ε, εισοδήματα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν θα πρέπει να υπάρξει ευθύ δαπάνη και των στρατιωτικών πόρων, συνδυασμό των στρατιωτικών δυνάμεων με τι αστυνομικέ, τι τελωνιακέ και να καλύπτουμε τι ανάγκε αντιμετώπιση τρομοκρατών και εγκληματιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Σμόκοβα. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σήμερα, σε περίοδο κρίσεων και ιδιαίτερων αναγκών, είναι φυσικό να έχουμε μικρότερα, λιγότερα κονδύλια για τον αμυντικό τομέα. Γι' αυτό χρειάζεται καλύτερο συντονισμό και σχεδιασμό στον αμυντικό τομέα, ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο έργο που θα επιτελούμε και να αποφύγουμε επικαλύψεις έργου σε περιόδους ε, εξτρεμιστικές ακραίων θέσεων και ξενοφοβίας η κοινή πολιτική άμυνας είναι πολύ σημαντικότερη από ό,τι οποτεδήποτε στο παρελθόν εκφράζομαι υπέρ της ε, κοινή αμυντικής πολιτικής, αλλά και για ένα κοινό συντονισμό και κοινό έλεγχο των επιμέρους συνιστοσών αυτής της αμυντικής πρωτοβουλίας ώστε να αποφύγουμε κατάχρηση των πληροφοριών. Στην χώρα μου είχαμε από πλευράς ε, στρατιωτικών υπηρεσιών κατάχρηση των δικαιωμάτων τους με παρακολούθηση των συνομιλιών και συνδιαλέξεων των πολιτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος αγορητής, κυρία Μπιλμπάο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Άστον, μεταξύ στα όσα αναφέρατε, για, αναφέρατε και την βελτίωση του σχεδιασμού για την αποτελεσματικότητα στις δράσεις μας στο κέρας της Αφρικής. Στον ε, Ινδικό ωκεανό έχουμε τον στόλο που αλλιεύει ε, τόνο από πλευρά τη Ισπανία και, ε, και των Βάσκων. Αυτά τα σκάφη υφίστανται επιθέσει των πειρατών και βρίσκονται υπό την προστασία τη δράση Αταλάντη που είχε οδηγήσει και σε ψήφισμα την Ευρωβουλή πέρυσι. Υπάρχουν τώρα προβλήματα διότι δεν μπορούν να εξοπλιστούν αυτά τα πλοία με βαρύ οπλισμό ώστε να προστατεύονται καλύτερα γιατί δεν δίνουν αυτή την άδεια οι αφρικανικές αρχές των αφρικανικών κρατών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι επετεύχθη για να βελτιωθεί η ασφάλεια στα σκάφη που αλλιεύουν ε, βασκικά και ισπανικά τον τόνο στον Ινδικό ωκεανό σε σχέση με τα όσα αναφέρατε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Ο επόμενος ο κύριος Τρεμόπουλος. Ένα λεπτό παρακαλώ κύριε Τρεμόπουλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω την ε, κυρία Άστον για τη μυστική συμφωνία που έχει αποκαλυφθεί στην εφημερίδα new europe μεταξύ παπανδρέου μέρκελ και σαρκοζή για την αγορά γερμανικών και γαλλικών όπλων αξίας δέκα εκατομμυρίων ως όρο για την χορήγηση του νέου πακέτου βοήθειας. βεβαίως η κυρία άστον δεν ακούει αυτή τη στιγμή αλλά θα ήθελα να μου σχολιάσει αυτή ακριβώς την ε, είδηση από μια έγκυρη εφημερίδα την ίδια στιγμή που υπάρχουν αντικοινωνικέ περικοπές στον προπολογισμό για το 2012 και ε, την ίδια στιγμή τα εξοπλιστικά ε, προγράμματα αυξάνονται κατά 18,2% και οι δαπάνε υπέρ του νάτο κατά 50%. Πρόκειται αν αληθεύει για ένα ευρωπαϊκό σκάνδαλο με τεράστια σημασία και γιατί τα κόμματα που κυβερνούν σήμερα στην ελλάδα εμπλέκονται αλλά και γιατί υπάρχουν μίζες τόσα χρόνια από γερμανικές και άλλες εταιρείες. θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν συμφωνεί η κυρία άστον με τον εξαναγκασμό της ελληνικής κυβέρνησης στο να συνεχίσει αυτή τη διπλωματία των εξοπλισμών και αν μπορεί να μας βοηθήσει τη χώρα δηλαδή για να απελευθερωθούμε από τα εκρεμή ζητήματα που ε, υπάρχουν με την τουρκία αντί να παρακολουθεί να βουλιάζουμε ακόμη περισσότερο στην κρίση. Ευχαριστούμε. Κυρία Φερέιρα. Ο κύριος Φερέιρα, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Εδώ πρέπει να δούμε το βασικό θέμα της συζήτηση που γίνεται. Υπάρχουν κάποιοι που μιλούν για την ε, περικοπή δαπανών, για τους φτωχούς και εργαζομένους της Ευρώπης και εντοπίζουν βέβαια το πρόβλημά τους στο δημοσιονομικό έλλειμμα και όχι στους ανθρώπους και στους περιορισμούς τους μισθούς ε, που πλήττουν ε, τις πολιτικές κοινωνικής προστασίας, τις κοινωνικές πολιτικές γενικότερα και την εκπαιδευτική πολιτική. Αλλά χωρίς περιστροφές λένε ότι πρέπει να προασπιστούμε τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να επηρεαστούν αυτές από τις περικοπές στον προπολογισμό ζητούν νέα όθηση σε αυτέ τι δαπάνε και τα κονδύλια. Όπω μα είπε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, νέα όθηση στην συνεργασία με τον ΝΑΤΟ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα, το συνδυασμό των ε, στατιωτικών μα επιχειρήσεων και τη βιομηχανία ε, του πολέμου. Δηλαδή, μιλάμε για νέε εκστρατείε που ετοιμάζονται και για μια επικίνδυνη τάση να παραμείνει η, κρίση και σε αυτό το τομέα. Οι αντικοινωνικέ πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ο αγώνα για την ειρήνη πρέπει να πηγαίνουν πηγαίνουν μαζί. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε. Στη συνέχεια, Σίνκλερ. Η κυρία Σίνκλερ έχει τον λόγο. Uh, Σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε όταν οι χώρες μας, για τις χώρες μας αναφέρονται αυτά στο σώμα και έχουμε το θέμα των στρατιωτικών δυνάμεων και το χρησιμοποιούμε στον πληθυντικό, τις στρατιωτικές μας δυνάμεις. Ε, δυνάμεις ε, στο Αφγανιστάν κάνουν εξαιρετική δουλειά από ό,τι μπορέσαμε να διαπιστώσουμε και προσωπικά. Είναι οι φορολογούμενοι του Ηνωμένου Βασιλείου που διαθέτουν τους περισσότερους στρατιώτες, όχι άλλες ευρωπαϊκές χώρες ε, και Κανένα μέλος της Ευρωβουλής δεν έχει δικαίωμα να περιγράφει αυτές τις δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου ή άλλες ως δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπηρετούν την, ε, αυτής μεγαλειότητα οι δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, την Βασίλισσα της Αγγλίας ε, και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αν δεν υπάρχει ομοφωνία στο ευρώ, πώς είναι δυνατόν για τέτοια θέματα αμυντικά να υπάρξει ομοφωνία. Και έχουμε και ένα πρόβλημα, δηλαδή σε σχέση με την, το, την πρώην ιδιότητα ε, από πλευράς της S&D, της ομάδας αυτής ως ταμεία τι, πώς μπορείτε εσείς να είσαστε αντικειμενικοί για αυτά τα θέματα και σε σχέση με την ε, παρέμβαση που έγινε σε σχέση με τα πυρηνικά πώς είναι δυνατό να, να δεχθείτε κάτι τέτοιο ευχαριστώ σας ευχαριστώ στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο ο κύριος ε, ε, ευχαριστώ πρόεδρε κυρία, είπατε, εκπρόσωποι, είπατε Και πρέπει εδώ να αναφερθώ στην παρέμβαση της κοινή χρήσης δυναμικού και ικανοτήτων που δεν είναι λέει επιλογή αλλά αναγκαιότητα. Ο στρατιωτικός αμυντικός προϋπολογισμός είναι πολύ χαμηλός και πρέπει το δυναμικό να διασφαλιστεί μέσω συνεργασίας. Προσωμιωτές για παράδειγμα μπορούν εναλλάξει να χρησιμοποιούνται και μέχρι και 16, από 16 αεροπλάνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Το ΝΑΤΟ έχει δείξει τη σωστή πορεία σε σχέση με αυτόν τον τομέα και για τις εναερίες μεταφορές. Κάθε χώρα καλύπτει με, τις δαπα... με τα κονδύλια της ένα συγκεκριμένο αριθμό πτήσεων. Και έχουμε και τη συνεργασία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας. Το ένα κράτος διαθέτει για παράδειγμα τις βάσεις, το άλλο τις στρατιωτικές δυνάμεις και εξοπλισμό. Και όσον αφορά την βελτιστοποίηση του δυναμικού και των δυνατοτήτων μας μέσω μεταφοράς ε, ε, ικανότητας. Αυτό το πρότυπο πρέπει και σε άλλους τομείς να μπορέσει να επεκταθεί και να χρησιμοποιηθεί στην λειτουργικότητα και στην υποστήριξη επιμελητιακά, π.χ. ελικόπτερα ή ε, όσον αφορά κανονιοφόρους ε, ε σκάφη που κάνουν ναυτικές περιπολίες. Σας ευχαριστώ. Στο τέλος θα λάβει τον λόγο ο κύριος Σκίνερ τελευταίος παρακαλώ. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή. Αφού πέφτει ε, το ποσοστό του ΕΠ θα πέσει ε, και ο αμυντικός υπολογισμό. Ε, πρέπει να το συνηθίσουμε. Και όλες αυτές οι περικοπές ουσιαστικά σπρώχνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια αμυντική παγίδα. Δεν θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές και μελλοντικέ δεσμεύσεις. Τι θα πρέπει να κάνουμε δεν μπορούν βιομηχανικά να εργαστούν μόνο τους τα χάρη, τα κράτη, οι προμήθειες, τεχνολογίες, όλα αυτά θα πρέπει να μπουν σε ένα ε, κοινό κορβανά και να είναι διαθέσιμο το δυναμικό για όλους. Νομίζω ότι έχουμε ευθύνη να ε, διατηρήσουμε το συντονισμό της κοινή πολιτικής ασφαλείας. Άκουσα κάποιους από τους προλαλήσαντες, από τον κύριο Βανόρντα παραδείγματος χάρη, να μιλά για το ΝΑΤΟ. Ε, η άποψή του δεν είναι σωστή και αυτό που λέει για τους γραφειοκράτες δεν κατάλαβα τίποτα. Τι εννοεί. Δεν θέλετε και εσείς να έχετε το γραφείο σας κύριε Βανόρντεν και το προσωπικό σας στις Βρυξέλλες. Α, και αυτό γραφειοκρατικό δεν είναι εκτός εάν ε, διάβασα λάθος τα στοιχεία. Πριν ασκείτε κριτική, καλύτερα διορθώστε τα του οίκου σας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο να δώσουμε το λόγο σε άλλους συναδέλφους στη διαδικασία Catch the Eye. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή κύριο Λίζε για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος για να κερδίσουμε χρόνο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους σε σχέση με την εκθεσή μου. Και τα θετικά σχόλια, αλλά και τις κριτικές. Ε, ουδής τέλειος. Εάν ε, όλα τα σχόλια αυτά, όλες τις παρατηρήσεις ε, τις χρησιμοποιούσα, θα μπορούσα να γράψω μια καινούργια έκθεση Ακούστηκα πολλά ενδιαφέροντα σε σχέση και με την αμυντική πολιτική της Ευρώπης. Συνειδητοποιώ βέβαια ότι η έκθεσή μου δεν πρόκειται να λύσει όλα τα προβλήματα. Η μόνη μου πρόθεση ήταν να επισημάνω ορισμένα βασικά ζητήματα στο πλαίσιο και της ε, τρέχουσας ε, χρηματοοικονομικής κρίσης. Να δω δηλαδή την κρίση υπό το πρίσμα της άμυνας. Και να εντοπίσω ποιε είναι οι απειλέ, ποιε είναι οι ευκαιρίε. Χαίρομαι πολύ που οι περισσότεροι από εσάς υποστηρίζετε τον πυρήνα της έκθεσής μου. Βέβαια δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε την άμυνα, Αυτό είναι το, αυτή είναι η ουσία της έκθεσης. Αλλά πολλοί ε, μπορούν να διερωτηθούν πού απευθύνεται αυτή η έκθεση τελικά. Εγώ δεν νομίζω ότι το βασικό μήνυμα η βασική έκθεση απευθύνεται στην ε, κυρία Άστον, που βέβαια έχει στηρίξει τα περισσότερα μηνύματά μας. Νομίζω ότι απευθύνεται περισσότερο στα κράτη-μέλη, στα εθνικά κοινοβούλια αυτή η έκθεση. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει με τις κυβερνήσεις να έχουμε διάλογο όταν βέβαια εγκριθεί αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Απάντησε τόσο γρήγορα ο κύριος Λίσεκ που ξέχασα, δεν πρόλαβα μάλλον να ρωτήσω τον κύριο Σκίνερ αν δεχόταν την ε, μπλε κάρτα από τον κύριο Βανόρντεν. Λοιπόν, κύριε Βανόρντεν, θέλω να απαντήσω στον αγαπητό φίλο και συνάδελφο Σκίνερ ε, σε αυτό που είπε. 30 χρόνια ήμουν, ξέρετε, στρατιωτικός ε, ε, στις ένοπλες δυνάμεις του στέματος και έχω πάει σε πολλά, ε, σε πολλά μέρη του κόσμου και όταν έφυγα στο στρατό και ασχολήθηκα με την πολιτική και περίμενα να έχω ένα έδρανο, για λίγο χρόνο ήμουν και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκεί είδα από μέσα το πώς εργάζεται η Κομισιόν. Αυτά όλα μου έδωσαν ε, και την εμπειρία μου για να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου ως βουλευτή σήμερα. Θέλω τώρα να δώσω το λόγο στην είπατε εκπρόσωπο την κυρία Άστον. Σας παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much, Mr. Well, um, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και άκρο σημαντική συζήτηση και αυτό κυρίως γιατί βλέποντας ε, την οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν ε, τα κράτη-μέλη αλλά και οι διάφοροι οργανισμοί και τα θεσμικά όργανα είναι πραγματικά ζωτική σημασία να συζητήσουμε το πώς μπορούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να ανταποκριθούμε ε, στην κρίση και στις απειλές ασφάλειας που αντιμετωπίζουμε είτε ως μεμονωμένα κράτη είτε ως βουλευτές είτε ως θεσμικά όργανα. Και Νομίζω ότι κανένας δεν θα εκπλαγεί ε, εάν πω ότι αυτές οι συζητήσεις είναι συζητήσεις που έχω συνέχεια σε τακτά διαστήματα με τον ε, κύριο Ράσμουσεν και όταν συμμετέχω με δικό του αίτημα ε, στις, στους σχηματισμούς τους, των εξωτερικών υποθέσεων και των αμυντικών θεμάτων στο ΝΑΤΟ. Και πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα ε, τι αποστολέ και επιχειρήσει που διεξάγουμε αυτή τη στιγμή και θέλουμε να δούμε πώ μπορούν να ε, έχουν την καλύτερη δυνατή συνεργασία και συμπλήρωση με άλλε επιχειρήσει και αποστολέ του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα όταν ε, συμπεριφέρθηκε όπως συμπεριφέρθηκε τον Αύγουστο του 8 η Ρωσία, είχαμε μια επιχείρηση στη Γεωργία. Εξακολουθούμε να έχουμε εκεί ε, προσωπικό για να είναι ασφαλή τα σύνορα, για να μπορεί επίσης ε, ο κόσμος να ζει κανονικά τη ζωή του. Επίσης, πολλοί μίλησαν για το κέρας της Αφρικής. Πραγματικά έχει γίνει καταπληκτικό έργο και συνεχίζει να γίνεται εκπληκτικό έργο από την επιχείρηση Αταλάντη και πολλά κράτη-μέλη ήταν πρόθυμα να συνεισφέρουν ε, σκάφη, ελικόπτερα ε, και εμπειρογνωσία. Οι Βρετανοί του Νόρθουτ βέβαια ε, και ο Βρετανός Ναύαρχος είναι αυτός ο οποίος έχει την, ε, αυτή τη στιγμή τη διοίκηση της επιχείρησης αλλά όλοι αυτοί καταβάλουν ε, σημαντικές προσπάθειες και για την λειτουργία του επισητιστικού προγράμματος γιατί ο κόσμος εκεί πραγματικά λιμοκτονεί και πρέπει να τους μοιραστούν τρόφιμα. Υπάρχουν επίσης απειλές ομοιρίας, Απειλεί επίσης για ε, τον τουρισμό. Είναι πολύ σοβαρά θέματα όλα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων. Όχι βέβαια να υποκαταστήσει το ΝΑΤΟ, αλλά να συνεργαστεί με το ΝΑΤΟ. Και ίσως το καλύτερο παράδειγμα που θα εξηγήσει όλα αυτά που λέω, είναι αυτό που γίνεται σήμερα στο κοσφοπέδιο. Η Γιούλεξ του κοσφοπεδίου είναι η λεγόμενη ε, δεύτερη ανταπόκριση, δευτερογενής ε, αντίδραση, όταν δηλαδή οι αξιωματούχοι μας προσπαθούν να σταματήσουν ε, κάποια κρούσματα βίας που βλέπουμε να εκδηλώνονται αυτή τη στιγμή. Συνεργαζόμαστε με τις νατοικές δυνάμεις και υπάρχει και η τρίτη μονάδα αντίδρασης. Είναι πολύ κίνδυνο, είναι πολλές οι δυσκολίες Είδαμε τι έγινε με Σερβία, μεταξύ Σερβία και Κωσυφοπέδιου. Πρέπει λοιπόν να δοθεί μια διεθνή απάντηση σε όλα αυτά. Και τα κράτη-μέλη όμω ελεύθερα πρόθυμα, τα ίδια εθελοντικά προσφέρονται να βοηθήσουν έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικά. Αστυνομική υποστήριξη για παράδειγμα. Όλα αυτά είναι διαφορετικά σε σχέση με αυτά που κάνει ο ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ συγγνώμη, όταν παρέχει στρατιωτική υποστήριξη. Νομίζω ότι όμω σε όλε αυτέ τι επιχειρήσει συνεργαζόμαστε πολύ στενά με το ΝΑΤΟ παράδειγμα, του χαρτών με τον ΝΑΤΟ συζητούσαμε πώ θα μπορούσαμε να στηρίξουμε ε, καλύτερα την επιχείρηση στη Λιβύη. Το ΝΑΤΟ είχε ε, επίγνωση τη κατάσταση, ότι δηλαδή είναι σε μια στρατιωτική επιχείρηση και άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να δουν ε, τι εξοπλισμό χρειάζεται για να υποστηριχθεί η παροχή τη ανθρωπιστική βοήθεια. Θέλω λοιπόν να πω σε όλου όσου ανησυχούν ότι υπάρχει αλληλεπικάλυψη, πρέπει να σα πω ότι και εμεί εργαζόμαστε σκληρά για να μην υπάρχει αυτή η αλληλεπικάλυψη εμείς ανταποκρινόμαστε όταν μας ζητά το ΝΑΤΟ ε, στήριξη. Δεν ε, χρειάζεται να σας θυμίσω αν ε, δείτε τι γίνεται σε χώρες που επιχειρούμε εκεί, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι ανησυχίας. Όταν συναντήθηκα με τους τέσσερις υπουργούς του Σαχέλ τις τελευταίες ημέρες, στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής προσέγγισης πρέπει να δούμε πώς θα τους στηρίξουμε διότι τους απασχολούν ε, οι τρομοκρατικές απειλές, μεταφορά όπλων από τη Λιβύη στο Σαχέλ, ε, ο υποσυτισμός ε, του πληθυσμού. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τους υποστηρίξουμε. Και κοιτάμε και το σκέλος της ασφαλείας. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας επίσης συνεργάζεται με το ΝΑΤΟ Παραδείγματος, ε, η εκρηκτικοί μηχανισμοί, η αυτοσχέδια εκρηκτική μηχανισμη είναι κάτι που απειλεί όχι μόνο το δικό μα προσωπικό, παραδείγματο χάρη στο Αφγανιστάν, ε, αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου. Και είναι ένα από τα θέματα. Αν μπορούμε λοιπόν να βρούμε ε, μια κοινή προσέγγιση, να δούμε πώ μπορεί να δημιούργησε να, ε, αυτούς τους ε, μηχανισμούς, δηλαδή την υπογραφή αν θέλετε που αφήνουν πίσω τους αυτοί οι εκρηκτικοί μηχανισμοί, οι διάφορες βόμβες. Αν μπορέσουμε και το κάνουμε αυτό θα σώσουμε ζωές σε όλο τον κόσμο. Και χρειαζόμαστε ανθρώπους που μπορούν να μας δώσουν απαραίτητη ε, εμπειρογνωμοσύνη. Και βέβαια έτσι θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το χρόνο, τα κονδύλια και τους πόρους μας. Επίσης για την κυβερνοασφάλεια πολύ σημαντικό και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Πρέπει να σας πω ότι με έχει προσεγγίσει ο Υπουργό Άμυνα ε, τον είπα για το θέμα αυτό, διότι μία από τις προκλήσεις ε, στην κυβερνοασφάλεια είναι ότι οι κυβερνοαπειλές δεν σταματούν στα σύνορα μιας χώρας και ξέρουμε ότι ε, οι ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις ε, που τέλος πάντων εννοώ ευρωπαϊκές ως ευρωπαϊκής ιδιοκτησίας επιχειρήσεις ή άλλες οντότητες που πλήττονται από αυτές τις κυβερνοεπιθέσεις και φυσικά και θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά και να τα αντιμετωπίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα επίσης να πω δύο πράγματα για να ολοκληρώσω. Πρώτα απ' όλα, Συμφωνώ με όλους όσους είπαν ότι πρέπει να είναι προληπτικό κατά κύριο λόγο το έργο μας. Η διαμεσολάβηση, η πρόληψη συγκρούσεων, η αξιοποίηση των πόρων μας για να αποτρέψουμε συγκρούσεις και προβλήματα. Πολύ σωστά. Αυτή είναι και η δική μας εστίαση και συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό επαναλαμβάνει είναι συμπληρωματικό σε ενέργειες που κάνουν άλλοι οι οποίοι εμπλέκονται στο, στα θέατρα επιχειρήσεων. Επίσης, πρέπει να είμαστε πραγματικά υπερήφανοι για ε, τους άνδρες και τις γυναίκες ε, που υπηρετούν, που, είναι, που έχουν αναπτυχθεί στα θέατρα επιχειρήσεων. Και πραγματικά υπηρετούν αυτοί οι άντρες, αυτές οι γυναίκες, ε, ιδίως στο Αφγανιστάν, με αυτοθυσία και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη για το έργο που κάνουν και πιστεύω ότι, και με βέβαια μάλλον ότι και εσείς οι βουλευτές το ίδιο πιστεύετε. Κυρία Ντότς μου κάνει επίσης μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, δηλαδή σε χώρες όπως είναι το Αφγανιστάν, αν μπορεί εκεί ε, να εξασφαλιστεί ε, η επιτυχία των δράσεων. Ο κύριος White συγκεκριμένα έχει κάνει πάρα πολύ καλά πράγματα στο Ιράκ. Αυτό ήθελα να τονίσω εγώ. Thank you very much, Vice Σας ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε Άστον. Και έτσι κλείνουμε την κοινή αυτή συζήτηση για την έκθεση του κυρίου Λίζεκ.